Καλημέρα σας. Ξεκινάμε κάπως καθυστερημένα. Θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, κυρία Υπουργό Τροφίμων Γεωργίας και Αλίας, ε, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, ε, η οποία θα μας παρουσιάσει τις προτεραιότητε της νέας εξάμενη Προεδρίας του Συμβουλίου. Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από μια παρουσίαση παραδοσιακή. Κυρίως γιατί είχαμε την ευκαιρία σήμερα το πρωί, μπορέσαμε να πάρουμε πρωινό μαζί της και την ευχαριστώ και υπάρχει μια σαφής δέσμευση ότι υπάρχει ένας μόνιμος ε, διάλογος ε, μεταξύ της Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι αυτή η αρχή είναι καταπληκτική. Κατόπιν ε, οι δραστηριότητε ε, στον τομέα της αλίας είναι πάρα πολλές, η ατζέντα είναι πάρα πολύ βεβαρημένη και φυσικά έχουμε πάρα πολλά θέματα να δούμε. Και το πρώτο θέμα είναι η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής εν εξελίξη. Είπαμε και στην κυρία Υπουργό ότι εργαζόμαστε για το θέμα αυτό. Είναι αλήθεια ότι ίσω δεν υπάρχουν επίσημε διαπραγματεύσει κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου τη Δανική Προεδρία. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε από την πλευρά της Προεδρίας ποια γραμμή ε, γίνονται οι συζητήσεις, ποια γραμμή ακολουθούν συζητήσεις ε, στους κόλπους του Συμβουλίου και πώς η ίδια η Προεδρία της Δανία έχει κατά νου να διευκολύνει τη διαδικασία για την επίτευξη της απαραίτητης συνένεση μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα. Εμείς ε, έχουμε κάποιες ανησυχίες ε, λόγω ε, της εμπλοκής στο Συμβούλιο για τα σχέδια διαχείρισης του Σαββριδού και της Ατζούγιας. Ξέρετε ότι ορισμένα κράτη-μέλη θέλουν να αγνοήσουν τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω ότι η Υπουργός την Καμισιόν ε, είπε την Επιτροπή ότι ε, πρέπει να έχουμε μια πραγματική συναπόφαση και θα πρέπει και το Συμβούλιο και η Επιτροπή να γνωρίζουν ε, και να έχουν πολύ ξεκάθαρο ποιες είναι οι ευθύνες του καθένα και οι αρμοδιότητες του καθένα και επίσης ε, πρέπει να έχουν πολύ ξεκάθαρο και ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι αλήθεια ότι ανησυχούμε ιδιαίτερα και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις εξωτερικές πτυχές της ε, κοινή ελευθερικής πολιτικής. Ανησυχούμε με από τις ε, συμφωνίες ε, που είναι υπό εξέταση αυτή τη στιγμή. Ορισμένε, όπως είπαμε, υπό εξέταση αυτή τη στιγμή. Επίσης, έχει δοθεί πολύ σαφή εντολή από αυτό το Κοινοβούλιο για τη συμφωνία με το Μαρόκο και υπάρχουν και άλλες συμφωνίες που είναι υπό διεκπαιρέωση. Και εμείς αυτό που αναμένουμε και αυτή είναι η πρώτη μου ουσιαστικά παρέμβαση ως πρόεδρο αυτής της Επιτροπής, αυτό που αναμένουμε είναι να πιστούμε για ε, τους λόγους ε, που θα διέπουν αυτές τις συμφωνίες και ε, να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο εγκαίρως για όλα όσα συμβαίνουν. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να επιτρέπουμε να γνωρίζουμε το Κοινοβούλιο σε τέτοιε θεμελιώδει συμφωνίε. Εγώ είμαι ότι από την πλευρά της ε, προεδρία της Δανίας θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και δυστυχώ μέχρι σήμερα, και το είδαμε και πολύ πρόσφατα στην περίπτωση του Μαρόκου, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ε, και άλλα πολλά θέματα που θα πρέπει να προσεγγίσουμε χωρί ε, καμία αμφιβολία, αλλά εγώ προτιμώ να είναι οι ίδιοι οι συντονιστέ, τα μέλη αυτή τη Επιτροπή που το πράξουν αυτό και χωρίς ε, χρονοτριβή να δώσω το λόγο στην κυρία Υπουργό και την ευχαριστώ για αυτή την πρώτη συνάντηση που είχαμε και επίσης ε, να σας πω ότι θα ακολουθήσουμε τη συνήθεια διαδικασία, θα δώσουμε μετά την παρέμβασή σας το λόγο στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων για τρία περίπου λεπτά παρέμβασης και να μας πούν τι θεωρούν κατάλληλο και στη συνέχεια ε, στους βουλευτές που θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν ε, το λόγο για ένα λεπτό περίπου. Θα θέλουν να πάρουν το λόγο. Αυτά από μένα. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την εκλογή σας ε, ως Αντιπρόεδρο. Είσαστε νέος ε, στη θέση σας αυτή. Ε, είμαι και εγώ νέα ε, στην Προεδρία. Είχαμε μία πρώτη συνάντηση τη Δευτέρα στο Συμβούλιο για τη Γεωργία. Και καθότι είμαι τόσο νέα στη θέση αυτή, θα ήθελα να σας πω ότι περίμεναμε περίμενα με αγωνία και χαρά το εξάμεινο της Προεδρίας, διότι νομίζω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην στις ε, καλές σχέσεις ε, μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Και θα ήθελα ε, σαφώς να πω ότι συμφωνώ ότι η συναπόφαση είναι συναπόφαση. Θα πρέπει να συνομιλούμε. Μπορούμε να γράψουμε ιστορία. Διότι πρέπει μαζί να πετύχουμε τη μεταρρύθμιση στην Αλία. Αυτό δεν έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά θα το κάνουμε. Και σε αυτό θα επικεντρωθεί ο διάλογός μας, ε, στον, στη μεταρρύθμιση της αλληλείας για τη, προς όφελος ε, των, ε, των λαών, των ανθρώπων και των αποθεμάτων. Ε, είναι ε, τιμή και χαρά μου να μιλήσω σήμερα για τις ε, προτεραιότητες της Δανέζικης Προεδρίας για το επόμενο εξάμεινο. Προσβλέπουμε στην επικοδομητική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Εγώ θα εκπροσωπώ τα 27 κράτη-μέλη του Συμβουλίου και είμαι αποφασισμένη να συνεργαστώ στενά μαζί σα. Πρώτα θα σα κάνω μια σύντομη εισαγωγή των βασικών προτεραιοτήτων τη Προεδρία. Θέλουμε υπεύθυνη, δυναμική, πράσινη και ασφαλή Ευρώπη. Θέλουμε να ετοιμάσουμε την Ευρώπη για το μέλλον από οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πλευράς. Η Δανέζικη Προεδρία θα ε, θέσει ε, ε, ένα προορατικό θεματολόγιο για πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε ανάπτυξη χωρίς να αυξήσουμε την ε, κατανάλωση ενέργειας ε, και άλλων πόρων. Και κάτι τέτοιο είναι δυνατόν. Η Προεδρία θα είναι φιλόδοξη και ρεαλιστική. Η πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη θα πετύχει μόνο εάν υπάρχει απαραίτητη υποστήριξη από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν, υιοθετηθούν οι προτάσεις και μεταφερθούν στην πράξη, δεν αρκεί να τις μεταφράσουμε σε διάφορες ε, ε, γλώσσες, θα πρέπει να τις ε, κάνουμε πραγματικότητα προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Το να επικεντρωθούμε στην πράσινη ανάπτυξη μας παρέχει και κάποιες ευκαιρίες. Ένα απλό και ευέλικτο πλαίσιο πράσινης ανάπτυξης ε, μπορεί να αποτελέσει ε, κίνητρο για καινοτομία και να δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, πετύχει ηγετική θέση στον κόσμο σε τεχνολογικούς τομείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στα χέρια της την ευκαιρία να δημιουργήσει πράσινη και οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη. Η κοινή αληθική πολιτική είναι ο τέλειος τομέας για να δοκιμάσουμε το όραμά μας ε, της πράσινης ανάπτυξης. Ε, είναι ένας από τους τομείς όπου η οικονομία εξαρτάται περισσότερο από το περιβάλλον και αυτό είναι το πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Θέλουμε η αλληλεία να ενσωματωθεί στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία της μεταρρύθμισης τη κοινή ε, αλληλευτική πολιτική για να ε, προχωρήσουμε προ αυτή τη νέα κατεύθυνση. Η νέα πολιτική θα πρέπει να διασφαλίζει την ε, βιώσιμη διαχείριση των αλληλευτικών πόρων, την προστασία των οικοσυστημάτων των ωκεανών μας και το συμφέρον όλων μας ως καταναλωτές και πολίτες και φορολογούμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ασχοληθούμε με τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερική πολιτικής ε, στο Συμβούλιο ε, του Μαρτίου, του Απριλίου, του Μαΐου με στόχο να πετύχουμε μια γενική προσέγγιση τον Ιούνιο, κάτι που θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί σας εδώ στο Κοινοβούλιο ε, στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Η μεταρρύθμιση αυτή έχει πολλέ πτυχέ και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρεις από αυτέ. Ε, η πρώτη έχει να κάνει με τις απορρίψεις. Πρέπει να εργαστούμε ώστε να αποφύγουμε τα ανεπιθύμητα αλλιεύματα και ουσιαστικά να δώσουμε τέλο ε, στην πρακτική των απορρίψεων. Από τη μία μεριά λέμε ότι δεν υπάρχουν ε, αρκετά ψάρια για όλους τους αλληλείς, από την άλλη οι αλληλείς μπορούν να ξαναδείχνουν τα αλλιεύματά τους στη θάλασσα. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Οι άνθρωποι της Ευρώπης ε, δεν το θέλουν αυτό. Αυτό αποτελεί σπατάλη τροφής και θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να λυθεί το πρόβλημα των απορρίψεων, αλλά πραγματικά πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια. Ας συνεχίσουμε τις εργασίες ε, στα πλαίσια αυτής της πρότασης για μεταρρύθμιση. Ε, έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Ε, το πρόγραμμα για τις ε, πλήρως τεκμηριωμένες, για την πλήρως τεκμηριωμένη αλλήλεια είναι ένα καλό ξεκίνημα. Το δεύτερο, η δεύτερη πτυχή που θα ήθελα να αναφέρω είναι η περιφερειοποίηση και η αποκέντρωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της μεταρρύθμισης. Φαίνεται να έχουμε μια καποστολή εικόνα του πού θέλουμε να πάμε και τι ακριβώς θέλουμε. Ξέρω ότι αυτό το θέμα ε, ενδιαφέρει πολλούς από εσά και ότι πολλοί απογοητευτήκατε με το πεδίο εφαρμογή της πρότασης. Ας ε, εργαστούμε σκληρά, ας ε, καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη και πρακτική και εφικτή πρόταση. Ε, θέλουμε πολύ να ακούσουμε τις ε, απόψει σα για το θέμα αυτό ε, και περιμένουμε τα αποτελέσματα της ακρόασης του Μαρτίου. Η τρίτη πτυχή είναι τα TFC, οι μεταβιβάσιμες αλληλευτικές παραχωρήσεις. Μερικοί θεωρούν ότι αυτό αποτελεί ιδιωτικοποίηση της θάλασσας ή πιστεύουν ότι αντίκειται στο στην ιδέα των κοινών αγαθών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, εργαστούμε εντατικά στο σημείο αυτό της μεταρρύθμισης ε, για να βρούμε ε, κάποια κοινή κατανόηση. Προσβλέπω στην ακρόαση που θα κάνετε τον Απρίλιο και θέλω πολύ να ακούσω τα αποτελέσματα των συζητήσεών σας. Θα ήθελα επίσης να δράξω την ευκαιρία να αναφερθώ στα μακροπρόθεσμα προγράμματα διαχείρισης προτού επανέλθω σε, άλλα, σε άλλες πτυχές του πακέτου μεταρρύθμισης. Ε, η μακροπρόθεσμη διαχείριση βρισκόταν στην καρδιά του πακέτου μεταρρύθμισης του 2002 καθώς και του παρόντος. Ωστόσο, πρέπει ε, εκ νέου να ε, καθορίσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για μακροπρόθεσμη διαχείριση στα πλαίσια της ε, νέας ε, συνθήκης. Αυτό το θέμα είναι πολύπλοκο και η Προεδρία ελπίζει να μπορεί να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί όλα τα θεσμικά όργανα. Η πρόταση για νέα κοινή οργάνωση αγοράς στόχο έχει να στηρίξει τους γενικούς στόχους της μεταρρύθμισης. Θα πρέπει να εστιάσουμε στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ε, των ε, ευρωπαϊκών προϊόντων αλληλείας, ε, εστιάζοντας ταυτόχρονα στα βιώσιμα προϊόντα. Τη στιγμή που οι πόροι είναι ελάχιστοι και υπάρχει τεράστια εισαγωγή ε, ψαριών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες ε, φαίνεται λάθος να αποσύρουμε μια πολύ καλά ψάρια από την αγορά με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα λήξει με την πρόταση της Κομισιόν και οι Υπουργοί θα έχουν μια σχετική συζήτηση τον Μάρτιο. Το άλλο σημαντικό θέμα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, ε, Θάλασσας ε, και Αλληλείας. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να βρούμε τους, τα αντικείμενα που, τους τομείς που θα αποτελέσουν αντικείμενα τη χρηματοδότησης. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στις περιβαλλοντικές στοιχεία, στην βιωσιμότητα και την καινοτομία. Αυτά δημιουργούν θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη κάτι που είναι απολύτω απαραίτητο στι ε, παράκτιε ε, κοινότητέ μας. Θα εργαστούμε σκληρά ώστε το Ταμείο αυτό να συνδυαστεί με τις άλλες νομοθετικές προτάσεις και θα έχουμε ε, έναν, μια συζήτηση γενικού προσανατολισμού πριν το, κατά, το Συμβούλιο του Μαρτίου προτού στοχεύσουμε στην, σε κάποια μερική γενική προσέγγιση τον Ιούνιο. Τέλος, ε, θέλω να ε, τονίσω ότι ε, η Δανέζικη Προεδρία χρειάζεται την βοήθεια και υποστήριξή σας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε καλή και στενή συνεργασία μαζί σας για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα και επιτρέψτε μου σύντομα να παρουσιάσω τις θέσεις της Προεδρίας για, άλλα, για άλλους φακέλους, για άλλα θέματα που ήδη συζητιώνται ε, στα θεσμικά μας όργανα ή προτάσεις που πιθανότατα ε, θα υποβάλει η Κομισιόν τους επόμενους μήνες. Ε, ξεκινώ με την τροπολογία του κανονισμού για την αλία βαθέων υδάτων που υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας Δανέζικης Προεδρίας το 2002. Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα για πολλούς από τους εταίρους μας στον Ατλαντικό Ατλαντικό, στα Δυτικά ύδατα και ε, θα το συζητήσουμε αυτό μόλι η Κομισιόν υποβάλει την πρότασή σα. Επίση θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας ε, για το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα διαχείρισης ε, για τον Σολομό τη Βαλτική, καθώ και άλλε προτάσει. Και τέλο, κύριε Πρόεδρε, φτάνω στο, στην εξωτερική διάσταση τη πολιτική αλίας μα το, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η ε, οι συμφωνίες εταιρικής, ε, οι αλληλευτικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης ε, πρέπει να είναι περιβαλλοντικές, οικονομικά βιώσιμες και να σέβονται το διεθνές δίκαιο. Βούμε, όπως προτείνει η Κομισιόν, ότι είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε τις βασικές αρχές της εξωτερικής διάστασης στον βασικό κανονισμό. Επίσης, σημαντικό είναι να αναφέρεται ρητά ότι η εξωτερική διάσταση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής θα ακολουθεί ε, τις ίδιες αρχές και τα ίδια πρότυπα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα πιο σημαντικό, η ε, αλληλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών θα πρέπει να γίνεται μόνο όπου υπάρχουν πλεονάσματα από θεμάτων. Καλύτερη επιστημονική συμβουλή, καλύτερος έλεγχος ε, είναι πολύ σημαντικά θέματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε. Και τέλος, οι συμφωνίες θα πρέπει να ωφελούν και τις τρίτες χώρες, όπως άλλωστε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος μας είναι να υιοθετήσουμε ε, συμπέρασματα του Συμβουλίου για την εξωτερική διάσταση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής κατά το Συμβουλίο του Μαρτίου. Υποθέτω ότι πιο πολύ προσοχή θα δοθεί στο Μαρόκο. Η Κομισιόν έχει υποβάλει τη σύστασή της για διαπραγματευτική εντολή για νέο πρωτόκολλο. Με την πρώτη ματιά αυτό φαίνεται να προχωράει προς τη σωστή κατεύθυνση και να έχει, να γίνει πιο σφιχτή η συμφωνία αυτή ε, και να ε, έχουν ληφθεί υπόψη οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί και μεταξύ άλλων και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας ε, διαβεβαιώσω ότι η Δανέσκη Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια τους προσεχείς μήνες για να έχουμε καλό διάλογο ανάμεσα στα θεσμικά μας όργανα. Θα κλείσω την παρουσίαση αυτή ε, αναφέροντας ότι ο τίτλος, το σύνθημα ε, του προγράμματος της Δανέσκης Προεδρίας είναι «Η Ευρώπη εργάζεται». Και Και δεν μιλάμε μόνο για όλους τους άλλους. Και εμείς θα εργαστούμε πολύ σκληρά για να διασφαλίσουμε βιώσιμο μέλλον για τους αλληλείς μας και για τα αλληλευτικά μας αποθέματα. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία μαζί σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Υπουργό. Να ξεκινήσουμε με τις παρεμβάσεις των διάφορων συντονιστών. Έχουμε εννέα άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο. Έτσι λοιπόν για να μπορεί να απαντήσει και η κυρία Υπουργό, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι, να σεβαστείτε δύο λεπτά οι συντονιστέ και ένα λεπτό οι υπόλοιποι. Εξ του ΕΛ και κυρία Φράγκα, καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την κυρία Υπουργό. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα θέματα. Το ένα είναι θεσμικό και νομίζω ότι εδώ έχουμε σοβαρή σύγκρουση με το Συμβούλιο από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα και τα δύο σημεία κλειδιά ήταν, όπω είπε ο Πρόεδρος στα σχέδια διαχείρισης όπου το Συμβούλιο ε, αρνείται συνεχώς να δεκτεί το Κοινοβούλιο να μπορεί ε, να γνωμοδοτήσει για το θέμα του Harvest Rule και το άρθρο 43.3 ε, για την αποκλειστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου για τον καθορισμό τάκνη ποσοστώσεων δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει το Συμβουλίο ό,τι θέλει όπως λέει ο βασικός κανονισμός. Αυτό είναι απαράδεκτο και εσείς μπλοκάρετε πάρετε κάποια σχέδια διαχείριση που ο ίδιο ο κλάδο ζητά να ρυθμιστεί το θέμα αυτό διαπαντό. Δεύτερο, θέμα διεθνού πολιτική. Εσείς ε, συνεχώς είστε αντίθετοι στη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνεδριάση συντονισμού, όχι διαπραγμάτευσης, γιατί η διαπραγμάτευση είναι ε, πραγματικά αποκλειστική αρμοδιότητα της Κομισιόν, όμως αρνείστε να συμμετάσχει το Κοινοβούλιο όπως συμμετέχει και το Συμβούλιο στις διεθνείς συνεδριάσεις και στις διμερείς συμφωνίες όπως ε, και στις περιφερειακές οργανώσεις αλίας και λέω ότι αυτό δεν σέβεται το πνεύμα ε, τη συνθήκη τη Λισαβόνα και θα αναγκάσετε το Κοινοβούλιο στο μέλλον να λάβει πιο δραστικά μέτρα, αν συνεχίσετε να αρνείτε. Δεν το λέω σε εσά ε, ε, προσωπικά, αλλά σα το λέω επειδή εκπροσωπείτε το Συμβούλιο και για το θέμα τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΛΠ. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να εγκριθεί αυτή η μεταρρύθμιση ε, υπό τη δική σας προεδρία, αλλά γιατί τις απορρίψεις ε, αυτό που είναι απαραίτητο είναι να αλλάξουμε το μοντέλο διαχείρισης όπως γνωρίζετε. Αν έχουμε απορρίψεις είναι γιατί έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης τα και ποσοστώσεων που ευνοεί τις απορρίψεις. Έτσι λοιπόν πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί στο θέμα αυτό και πρέπει να αλλάξουμε το θέμα διαχείρισης για την περιφερειοποίηση θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν γιατί η Κομισιόν τίποτα δεν παρουσίασε που να είναι περιφερειοποίηση αλλά το αντίθετο και το θέμα της ουσίας ε, εδώ ε, είναι θέμα αυτό ουσιαστικό ή θα έχουμε μία μεταρρύθμιση που θα είναι και οικονομικά βιώσιμη για το τομέα ή για το ταμείο θα πρέπει ε, να επανέλθουμε ε, στις επιδοτήσεις. Εγώ είμαι κατά του να δίνονται επιδοτήσεις στο στόλο, όμως νομίζω ότι πρέπει να τροποποιηθεί ο βασικός κανονισμός και να έχουμε ένα μοντέλο διαχείρισης ε, που να ε, είναι πέρα από αηφόρο περιβαλλοντικά, να είναι και βιώσιμο οικονομικά για τον τομέα. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην τροποποιήσουμε το μοντέλο της διαχείρισης. Νομίζω ότι είναι ζωτικό λοιπόν αυτό το θέμα για το Μαρόκο. Αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να το θίξω, θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς ε, έχετε την εντολή, συζητείτε στο Συμβούλιο, αλλά διαγράψατε, ε, καταργήσατε την αλή από το Φεβρουάριο και καθώς το Φεβρουάριο δεν θα υπάρχει Συμβούλιο Αλίας, πότε σκοπεύετε να το δείτε το θέμα αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που γνωρίζετε και τι θέλω να μου πείτε, πότε εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει σύμφωνα ή εντολή για τη διαπραγμάτευση. Ευχαριστούμε κυρία Φράγκα. Κύριε το για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρία Υπουργέ και εγώ σας καλωσορίζω και χαίρομαι που η Δανία ε, έχει τώρα την Προεδρία. Νομίζω θα συνεργαστούμε πολύ καλά. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια θέματα. Ε, έχετε ασχοληθεί και εσείς εντατικά με το θέμα. Το 2002 θέσαμε έναν υψηλό στόχο στο Johannesburg. Είπαμε ότι μέχρι το 2015 θέλουμε να περιορίσουμε την υπεραλίευση και να έχουμε ε, εφαρμόσει τα ε, σχετικά μέτρα μέχρι το 2015. Μέχρι τώρα βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Ε, καταρχήν ε, θέλουμε να ασχοληθούμε με το FMS και να δούμε πόσο ε, γρήγορα, ε, πόσο, πόσα μπορούμε να πετύχουμε μέχρι το 2015, διότι ως γνωστόν δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο αυτό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για μένα προσωπικά. Ε, θέλουμε να μειωθούν οι αλλιευτικές ευκαιρίες Ε, θα πρέπει όμως ε, να κοιτάξουμε και την κοινωνική πλευρά, όπως και την οικολογική, όπως είπε η κυρία Φράγα. Επίσης, να αναφερθώ στα ΤΑΚ. Είναι πολύ σημαντικό ότι στις διαπραγματεύσεις ε, είναι πολύ σημαντικό στις διαπραγματεύσεις να συμμετάσχει και αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, ε, είπατε ότι λείπουν πολλά επιστημονικά στοιχεία. Ε, νομίζω ότι πολλές φορές ε, τα κράτη-μέλη θελημένα εμποδίζουν την συλλογή στοιχείων. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις και επίσης ε, όσον αφορά την ε, απαγόρευση των απορρίψεων, πιστεύετε ότι αυτή θα πρέπει να ισχύει μόνο ε, για τα εμπορεύσιμα ή για όλα τα ψάρια. όσον Όσον αφορά τις ποσοστώσεις, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, έχουμε ένα ευέλικτο σύστημα. Μπορείτε να φανταστείτε ε, μεταφορά των ε, μη εξαντλημένων ποσοστώσεων από τη μια χρονιά στην άλλη. Γενικά, τι μορφή πιστεύετε ότι θα έχει ένα σύστημα ποσοστώσεων στο μέλλον. Γενικά, θα πρέπει να σκεφτούμε να μιλάμε όχι μόνο για απαγορεύσεις, αλλά και για κίνητρα και συστήματα αμοιβή. Ε, πιστεύουμε ότι ε, οι αλληλείς ε, που εφαρμόζουν κάποια νέα συστήματα θα πρέπει να αμείβονται. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν κάποια μέτρα ασφαλείας ώστε να μην έχουμε υπερβολική συγκέντρωση. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες εξαιρέσεις για τους μικρούς αλληλείς. Δεν σκέφτομαι όμως τους μικρούς όσον αφορά το μέγεθος των σκαφών, αλλά όσον αφορά ε, τον όγκο της αλληλείας. Ε, βλέπω ότι ο χρόνος μου τελειώνει. Ε, τελευταίο θέμα, το εξωτερική διάσταση, το Μαρόκο. Έχετε ένα ψήφισμα δικό μας. Στα πλαίσια της συνεργασίας θα ήθελα να αναγνωρίσετε ε, το ψήφισμα αυτό. Ε, η ομιλήτρια ζητεί ε, συγγνώμη από τους Γερμηνείς λόγω της φωνής της, επειδή είναι βραχνή. Μάλιστα, ο κύριος Γκαλκέρα από την Ομάδα Φιλελευθέρων και προσπαθήστε να είστε σύντομοι για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε, αλλά βέβαια δεν φταίει η Προεδρία. Κύριε Γκάλχερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο χειρότερος εχθρός μας είναι ο χρόνος, τελικά. Θα ακολουθήσω πάντως τις οδηγίες σας. Έχουμε την ευκαιρία σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι και άλλοι συνάδελφοι θα πρέπει να έχουν όμως την ευκαιρία αυτή να θέσουν ερωτήσεις. Η Υπουργός αναφέρθηκε σε κάποιες αλλαγές που υπάρχουν ανάμεσα σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές, στις, στη δυτική αν θέλετε θαλάσσια ζώνη. Μόνο και μόνο αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό επιχείρημα υπέρ της περιφερειοποίησης, υπέρ της αποκέντρωσης. Μιλήσαμε για τις απορρίψεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και τα απαραίτητα μέτρα διατήρησης, συντήρησης και θα πρέπει να δοθούν τα παρέτα κίντρα προ αυτό. Όσον αφορά τώρα την αλία μικρή κλίμακα. ουσιαστικά σκέφτομαι μικρά σκάφη τα οποία δεν, δεν ξεπερνούν καν την έκταση του Προεδρείου αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τους μικρούς αυτούς αλείς. Δεν είναι αυτά τα σκάφη τα οποία έχουν κάποια πολύ σημαντική επιζήμια επίπτωση όσον αφορά τα λευτικά αποθέματα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε λοιπόν με τους μικρούς αλείς. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διευθετήσει το ζήτημά τους. Θα ήθελα και εσείς όμως εκπροσωπώς στο Συμβούλιο να ασχοληθείτε με το ζήτημα αυτό. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει κάτι το οποίο συζητήσαμε συζήτησα και με τον συνάδελφο Chris Davis πριν από κάποιο καιρό και αναφέρομαι στους μικρούς λιμένες οι οποίοι είναι εντελώς κατακαιρματισμένοι ακριβώς επειδή η αλληλεία εκεί πέρα περιορίζεται όλο και περισσότερο. Ξέρετε εσείς ε, πολύ καλά πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει στα πλαίσια των κοινοτικών ταμείων να χρησιμοποιηθούν κάποιες χρηματοδοτήσεις, κάποια κονδύλια, προκειμένου να προσελκύσουμε επενδύσεις στους μικρούς αυτούς λιμένες, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες στους λιμένες αυτούς, προκειμένου να υπάρχει απαραίτητη υποδομή, προκειμένου να μπορούν να γίνουν επενδύσεις ε, στους λιμένες αυτούς. Δεν σας ζητώ να κάνουμε κάτι καινούριο. Ήδη οι φυσικοί πόροι υπάρχουν στους λιμένες αυτούς. Σας ζητώ απλώς να τους υποστηρίξουμε. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα διατήρησης, ε, μάλλον πιο συγκεκριμένα με συγχωρείτε όσον αφορά τις μεταβιβάσιμες ελευτικές παραχωρήσεις. Υπάρχουν χώρες που έχουν σημειώσει επιτυχία στον τομέα αυτό. Είναι όμως οι χώρες αυτές, μάλλον αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα καλά και σε άλλες χώρες. Αυτό μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα κινητοποιηθούν πιο γρήγορα, θα αγοράσουν όλες αυτές τις παραχωρήσεις και ουσιαστικά θα καταφέρουν να προσελκύσουν όλα τα αποθέματα, όλα τα ελιεύματα προς αυτές τις μεγάλες χώρες, προς δικούς τους λιμένες, προς δικές τους εταιρείες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν μέσω των TFCs να μην παραμερίσουμε τις μικρές χώρες. Όσον αφορά τους λιμένες, Ελπίζω ότι θα εργαστείτε μαζί μας και ότι η Προεδρία θα εργαστεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε τα πολιετή σχέδια διαχείρισης. Τα δυόμιση έτη τα οποία προβλέπονται δεν με ικανοποιούν. Η ανακοίνωση που έχουμε επιτάπητος αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο είναι μια ανακοίνωση που μας απασχολήσει, ιδίως το ζήτημα των κυρώσεων κατά τον χωρών αυτών που αλλιεύουν με μη βιώσιμο τρόπο. Ξέρω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα γενικό, θέλουμε όμως να προχωρήσουμε το ζήτημα αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτή μπορεί να επιφέρει κάποιες θετικές επιπτώσεις και αυτό, ελπίζω. Όλοι μας σήμερα έχουμε κάτι κοινό. Θέλουμε να αλλιεύουμε με βιώσιμο τρόπο Θέλουμε να προστατεύσουμε τα αποθέματα προκειμένου και οι μελλοντικέ γενέ να καταφέρουν να στηριχτούν στην αλία. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μάλλον έχω χάσει τη μάχη. Ε, ενώ σας ζητώ να είστε πιο σύντομοι, δεν το κάνετε, αλλά θα πρέπει να σας κόψω μάλλον τελικά. Δεν μου αρέσει, αλλά ξέρετε, ο χρόνο ε, τρέχει. Έτσι λοιπόν, ε, σα παρακαλώ προσπαθήστε. Εξ ονόματος των Πρασίνων, κυρία Λέβεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρα. Και θα ήθελα να καλωσορίσω την Δανέζα Υπουργό. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τις ε, προτεραιότητές σας και που έχετε αυτή την ολιστική προσέγγιση για το μέλλον της Ευρώπης ε, και ότι παρουσιάζεται τη υπευθυνότητα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η μεταρρύθμιση της κοινή ελευτική πολιτικής ε, και η συμπερίληψη της περιφερειοποίησης αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για να έχουμε μια νέα ολιστική προσέγγιση στις των θαλασσών μας και ξέρω ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν πολλές ερωτήσεις και φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει κάποιος ε, δισταγμός ε, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί η περιφερειοποίηση. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Υπουργών Ενέργειας Περιβάλλοντος και Γεωργίας για να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε μια πραγματικά περιφερειακή προσέγγιση με τη συμπεριλήψη και περιβαλλοντικής νομοθεσία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθούν στο να καταρτήσουν κάποιες κυρίες ε, αρχές για ε, κάποιους κανόνες για τον ε, έλεγχο της αλίας των αλευμάτων. Έτσι λοιπόν και τα περιφερειακά συμβούλια θα θέσουν θα, κάποια όρια, αλλά και σε πιο, τα πιο τεχνικά θέματα, όπως είναι οι μέρες στη θάλασσα και το μάτι του δικτύου, αυτά θα πρέπει να ρυθμίζονται σε τοπικό επίπεδο. Δεν θα ήθελα το Κοινοβούλιο να εμπλακεί σε ιδιαίτερα τεχνικές συζητήσεις. Νομίζω ότι δεν θα ήταν σωστή κατεύθυνση αυτή. Σε ό,τι αφορά στην εξωτερική διάσταση, Χάρηκα που άκουσα ότι θέλετε οι βέλτιστες αρχές να συμπεριλαμβάνονται στο βασικό κανονισμό. Νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστούμε για τη συμπερίληψη της ρήτρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλουμε να τονίσουμε και τη σημασία της διαφάνειας στα θέματα αυτά. Έχω και δύο ερωτήσεις. Ένα για τις μεταβάσεις βασιλευτικές περιχωρήσεις. Ένα ερώτημα. Έχετε ήδη τη σχετική εμπειρία. Είπατε στο πρωινό ότι θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικές, αλλά εθελοντικές. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά από την Αυστραλία Άκουσα ότι χρειάστηκαν τουλάχιστον 15 χρόνια για να το εφαρμόσουν αυτό, για να έχουν άτομα επί τους σκάφους. Ε, ε, τι λέτε εσείς, ποια είναι η αποψή σα για το χρονοδιάγραμμα που προτείνει Κομισιόν. Νομίζω ότι κινείται πολύ βιαστικά. Και τελευταία ερώτηση. ποιε είναι οι κυρίες προκλήσεις, οι κυρίες δυσκολίες που βλέπετε στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Θα μπορούσατε να τονίσετε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λομπάσεκ, ε, εκ του ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ επίσης, ε, κυρία Υπουργέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνετε σήμερα δυνατότητα να κάνουμε μία ανταλλαγή απόψεων. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις διαπραγματεύσεις σας. Κύριε Υπουργέ, η Δανία έχει τον μεγαλύτερο στόλο στη Βαλτική και έχει ειδικά δικαιώματα στα πλαίσια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Έχετε όμως και συγκεκριμένα καθήκοντα και ειδικέ υποχρεώσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που διεξάγεται στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθώ στα ζητήματα αυτά τα οποία ήδη αναφέρατε. Ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα άλλο από να συζητάμε τα ζητήματα αυτά συνεχώς στις συνεδριάσεις μας. Το ερώτημά μου λοιπόν έχει να κάνει κυρίως με τη ζώνη της Βαλτικής θάλασσας. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση όταν μιλάτε για περιφερειοποίηση. Πώς ακριβώς θα διεξαχθεί η περιφερειοποίηση. Τι κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσει. Ποιος θα πρέπει να είναι ο προσανατολισμός για την περιφερειοποίηση της Βαλτικής θάλασσας. Ποια στοιχεία θα πρέπει να περιέχει ποιες περιοχές θα πρέπει να αφορά. Και όταν, αφορά, όταν μιλάτε για απορρίψεις ή ανεπιθύμητα λιεύματα, πώς μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα αυτό συγκεκριμένα στη Βαλτική θάλασσα. Όταν λέτε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τις απορρίψεις, πώς αυτό θα πειράσει την παραγωγή. κάνετε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στα ποιοτικά νοπά αλλιεύματα σε σχέση με τα μεταποιημένα αλλιεύματα. Πώ θα εφαρμοστούν όλα αυτά στην Βαλτική θάλασσα και αναφέρομαι στη Βαλτική θάλασσα γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη ζώνη για την αλία. Επίσης, τι διαφοροποίηση θα γίνει ανάμεσα σε μεγάλους και μικρούς ελευτικού στόλου, Ποιο θα πάρει τι τελικέ αποφάσει, Ποια είναι η δική σα άποψη για τα ζητήματα αυτά. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, κυρία Υπουργέ, γιατί αναφερθήκατε στον Σολομό της Βαλτικής. Εγώ συντάσω μία έκθεση για διαφορετικά είδη αλίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αφορά που κάνετε, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε που σεβαστήκατε το χρόνο. Κύριος Φερέιρα, ξενόματος της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Δανικής Προεδρίας για την παρουσίασή της και για τη διαθεσιμότητά της να, συναντούμε, να συναντιόμαστε τους επόμενους 6 μήνες και να συζητούμε τα θέματα που έχουμε ενωπιών μας. Φυσικά το θέμα της μεταρρύθμισης είναι ένα μεγάλο θέμα. Εδώ εγώ θα ήθελα ε, να αναφερθώ στην ε, θέση της Δανίας ε, σε σχέση με τις μεταβάσιμες ελευτικές υπεραχωρήσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να απορριφθεί η πρόταση της Κομισιόν που είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να δώσουμε προαιρετικό χαρακτήρα σε αυτό το εργαλείο, έτσι δηλαδή κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει, ε, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του, αν θα πρέπει να θετήσει ένα τέτοιο σύστημα, αν θα εξυπηρετεί το στόλο του. Εγώ νομίζω ότι αυτή η θέση είναι πάρα πολύ σημαντική όταν προέρχεται από μια χώρα που έχει μάλιστα ίδια εμπειρία για την εφαρμογή αυτού του συστήματος και γνωρίζει τις συνέπειες της εφαρμογής του συστήματος Αυτό Έτσι λοιπόν εγώ θα ήθελα να προσδώσω δώσω αξία σε αυτή τη θέση. Επίσης ε, υπάρχει και ένα θέμα που θα τεθεί το επόμενο εξάμεινο και είναι το θέμα της, ε, των αλληλευτικών συμφωνιών, της ελευτικής συμφωνίας με το Μαρόκο. Εγώ θεωρώ καθώς ε, η Προεδρία γνωρίζει γιατί ε, το Κοινοβούλιο απέρριψε την παράταση της συμφωνίας, ε, υπάρχει και ένας λόγος πιο σημαντικός και για μας ο λόγος αυτός είναι ότι δεν σέβεται η συμφωνία αυτή το διεθνές δίκαιο. Και δεν ε, είναι μόνο ε, το ότι θα πρέπει να, χρησιμοποιηθούν ε, οι συμφωνίες αυτές υπέρ του συμφέροντος του λαού. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έγινε σεβαστό, μια προπόθεση που δεν έγινε σεβαστή στη συμφωνία που σύναψε η Κομισιόν και θα ήθελα να μου πείτε ποιοι μηχανισμοί προβλέπονται για να εγγυηθούμε αυτή τη φορά ότι και η βούληση του λαού της Δυτικής Αχάρας ε, πέρα από τα συμφέροντα του λαού θα λαμβάνονται υπόψη. Δηλαδή έχουμε τις μεροκινές αρχές να, λέμε, να λένε ποια είναι τα συμφέροντα του λαού της Δυτικής Αχάρας όμως υπάρχουν ε, νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού του λαού και εκπροσωπούνται στα Ηνωμένα Έθνη οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι λοιπόν αυτές οι αρχές ε, ε, έχουν, ε, μπορούν να τοποθετηθούν σχετικά και έχουν δηλώσει τη διαθεσιμότητά τους να διαπραγματευτούν μια συμφωνία. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Και να κλείσω με ένα σχόλιο. Εγώ πρόσεξα από την πλευρά της Δανικής Προεδρίας ε, κάποια ανησυχία στο να διαχωρίσει ε, τη Δανία ε, ως κράτος μέλος στο Συμβούλιο και το ρόλο της ως Προεδρία και θέλει να διατηρήσει μια ουδετερότητα. Εγώ θεωρώ ότι η ουσία των εκπεριτροπής Προεδριών είναι ακριβώ ότι το κάθε κράτος μέλος μπορεί να παρουσιάσει και να προωθήσει τις δικές του Θέσει κατά ένα εξάμεινο. Διαφορετικά δεν είχε κανένα νόημα αυτή η εκπεριτροπή προεδρία, γιατί θα μπορούσαμε να δώσουμε στον κύριο Φανροπόη ε, περισσότερο προσωπικό τεχοκνατών και θα μπορούσε αυτός να επιτελεί τις εργασίες. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να αναφερθείτε στη TFC και στην Ελευτική Συμφωνία με το Μαρόκο, σε αυτά τα δύο θέματα που έθεσα και ε, θα ήθελα ε, η Προεδρία της Δανίας ε, να υπερασπιστεί τις δικής της θέσεις κατά τη διάρκεια της άσκησης της Προεδρίας σας. Αυτή είναι η έννοια των Επιτροπής Προεδριών, όπως σας είπα. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Πριν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σαλαβράκο, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Καταρχήν, ε, να μας δώσει, κύριε Υπουργός, 10 λεπτά ακόμα, αν δύναται, για να έχουμε μια μεγαλύτερη συζήτηση και όταν ε, ε, πάρει το λόγο και ο τελευταίος συντονιστής να απαντήσει κυρία Υπουργό και κατόπιν ε, θα ε, δώσουμε το λόγο σε πέντε συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο αλλά για ένα λεπτό. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για τη γενοδορία σας. Ο κύριος Αλαβράκος τώρα. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ. θα είμαι σύντομος διότι όλοι όσοι προελάλησαν έδειξαν όλα ουσιαστικά τα θέματα. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος ε, Φεραίρα για το θέμα της ε, εκπεριτροπής προεδρίας. Εγώ πιστεύω ότι η εκπεριτροπής προεδρία δεν έχει ουσιαστικό ρόλο παρά μόνο δείχνει ότι τα κράτη-μέλη και η όλη Ένωση είμαστε δημοκρατικοί και το κυριότερο εποφελούμεθα την εμπειρία κάθε κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία εποφελείται της εμπειρίας των επιτροπών που συμμετέχουν όλοι οι υπόλοιποι και νομίζω ότι μεταφέρει αυτή την εμπειρία στην ε, εσωτερική διακυβέρνηση της χώρας του καθό μέρος θεωρεί ότι αυτή είναι σωστή. Συνεπώς από την Προεδρία τη δική σας περιμένω την ένδειξη της δημοκρατικότητας και εάν μπορείτε σε κάθε τομέα της δραστηριότητας να λάβετε υπόψη και την εμπειρία των επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θεωρώ ότι όλα τα θέματα τα οποία εθίχθησαν είναι ουσιαστικά. Σε εκείνο το οποίο θα έμενα είναι στο πώς θα ενισχύσουμε τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη με διαφορετικές πολιτικές να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν καλύτερες πρακτικές διότι οι αρμοδιότητες που θα εκορίζονται σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να είναι διαφορετικές και να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιομορφίες της κάθε περιοχής και εδώ έχουμε τη λεκάνη της Μεσογείου, τη λεκάνη της Βαλτικής και τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας οι οποίες έχουν διαφορετικές ιδιαιτερότητες η μια και πρέπει να προσαρμόσουμε μια γενικότερη πολιτική που να είναι σύμφωνη με τα δεδομένα των περιοχών αυτών. Σας εύχομαι και πάλι Καλή επιτυχία στην Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον όλων σας για τη συζήτηση αυτή. Θα ξεκινήσω απαντώντας στην ερώτηση για τα θεσμικά όργανα και την συνθήκη. Νομίζω ότι η συνθήκη είναι πολύ σαφής. Πρέπει να έχουμε συναπόφαση. Πρέπει να έχουμε κοινέ αποφάσεις ε, σχετικά με τη μεταρρύθμιση. Τόσο απλά. Οι, απο, ε, για τα τάκα και τις ε, ποσοστώσεις ε, ανήκουν στο Συμβούλιο, ενώ το πρόγραμμα διαχείριση αποτελεί αντικείμενο συναπόφασης. Ακούω όμως αυτά που λέτε. Μας λέτε ότι δεν συμμετέχετε αρκετά ότι δεν μπορείτε να συμμετέχετε στις ε, διαπραγματεύσεις για την εξωτερική πολιτική. Θέλετε να ενημερωνόσαστε όμως καλύτερα. Το σημειώνουμε. Θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι η πόρτα μας ανοιχτή. Η Δανέζικη Προεδρία είναι διατεθειμένη να έχει διάλογο ανα πάσα στιγμή. Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε την πόρτα μας λοιπόν, περάστε από την πόρτα μας αν χρειάζεται πληροφορίες. Υπήρξαν συζητήσεις σχετικά με το πώς είναι να είναι κανείς δανός, πώς είναι να είναι κανείς πρόεδρος, ε, πώς ε, είναι να κατέχει κανείς το ρόλο της Προεδρίας. Θα βγάλω λίγο το καπέλο της Προέδρου και θα σας πω ότι ήσασταν πολύ ευγενικοί και δεν μιλήσατε πολύ για τις εξωτερικές συζητήσεις για την Ισλανδία και τις Περόες Και μπορώ να καταστήσω απόλυτα σαφές ότι αντιλαμβάνομαι ότι η Δανία έχει ειδική σχέση με τις Φερόες νήσους και το ξέρετε αυτό όλοι. Οι διαπραγματεύσεις όμως για το σκουμπρί δεν είναι αντικείμενο της Προεδρίας, είναι διαπραγματεύσεις της Κομισιόν. και πραγματοποιούνται σήμερα. Δεν ε, μπορώ να σας ε, πω τίποτα για τα αποτελέσματα. Ε, μπορώ όμως να σας πω ότι θα είμαι πρόεδρος για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά λοιπόν τις κυρώσεις, θα θέσω τα θέματα προς συζήτηση. Δεν θα προσπαθήσω να κρύψω τίποτα κάτω από το τραπέζι. Θα θέσω το θέμα προς στο Συμβούλιο. Αντιλαμβάνομαι ότι ως Δανέζα αλλά και ως Πρόεδρος είναι σημαντικό να τα τονίσω αυτά, να ξέρετε ότι θα είμαι πιστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά με την νομοθετική ρύθμιση, νομίζω ότι είναι σημαντικό για όλους μας να καταλάβουμε Και κάποιοι από σας αναφέρθηκαν στη βιοπικιλότητα, στο Johannesburg, ε, τους στόχους του 2015 και τη βιωσιμότητα. Στα χέρια μας κρατάμε τη μελλοντική αλληλευτική πολιτική. Στα χέρια μας κρατάμε τη διαχείριση των αποθεμάτων. Και οφείλουμε στις μελλοντικές γενιές να προσέξουμε αυτά τα ε, πολύτιμα δώρα που μας δόθηκαν από τους ε, προγόνους μας και γι' αυτό αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό μιλώ για βιωσιμότητα. Αντιλαμβάνομαι ότι οι αλληλείς και οι, προσπα... οι αλληλευτικές ευκαιρίες βρίσκονται υποπίεση από... Ε, λόγω ένα σωρό προβλημάτων και τελικά όλα καταλήγουν στους αλληλείς. Η απάντηση όμως δεν είναι να πούμε στους αλληλείς κάντε ό,τι θέλετε. Η απάντηση είναι να βοηθήσουμε τους αλληλείς να έχουν διαφανή νομοθετική ρύθμιση η οποία να είναι και βιώσιμη. Ξέρω ότι σε πολλές χώρες ε, τα σκάφη κληρονομούνται από πατέρα σε γιο, όπως και το επάγγελμα. Και θα πρέπει στις επόμενες γενιές να μπορούμε να δώσουμε ε, αλληλευτικά αποθέματα ε, καθώς ε, και βιοπικιλότητα. Πώς θα το κάνουμε λοιπόν αυτό. Νομίζω ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική είναι αρκετά βιώσιμη όσον αφορά την προσέγγιση της στο, πρόγραμμα, στο πρόβλημα αυτό και την πρόκληση αυτή. Συμφωνώ με την κυρία Ρόντουστ που μιλάει για την ανάγκη για κίνητρα. Ε, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι η τηλεόραση κλειστού κυκλήματο, το CCTV και ο πλήρης έλεγχος των ε, αλλιευμάτων. Αυτό το έχουμε στη Δανία και φαίνεται να είναι χρήσιμο τρόπος να αποφύγουμε τις απορρίψεις. Πρέπει κάτι να κάνουμε για τις απορρίψεις. Αντιλαμβάνομαι ότι ότι αυτό δεν συζητιέται διότι πολλές χώρες ε, δεν ε, θέλουν ε, τηλεοράς του κυκλώματο στα σκάφη. Πρέπει να το συζητήσουμε όμως. Έχουμε πολλά προβλήματα, έχουμε πολλά πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Χρειαζόμαστε όμως και λύσεις. Η CCTV και η πλήρως τεκμηριωμένη αλία μπορεί να αποτελέσει μία από τις λύσεις. Όσον αφορά τις μεταβάσιμες αλλιευτικές παραχωρήσεις, τα TFC, Ε, να σας παρουσιάσω και εδώ τη θέση της Δανίας. Η θέση της Δανίας είναι ότι αυτό το δοκιμάσαμε. Ε, δεν μας πήρε 15 χρόνια η εφαρμογή, δύο χρόνια μας πήρε. Και καταφέραμε να έχουμε τέτοιου είδους ρύθμιση, χωρίς να έχουμε λιγότερα παράκτια σκάφη σε σχέση με τα άλλα σκάφη. Μπορεί να υπάρξει ισορροπία λοιπόν εντό ενό τέτοιου συστήματο. Αλλά να σα πω επίση ότι η θέση τη Δανία είναι ότι δεν κάνουμε σταυροφορία. Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι προαιρετικό για, χώρες, για τις χώρες. Αλλά ε, ως Προεδρία πρέπει να σας πω ότι ε, η πρόταση της Κομισιόν είναι να είναι υποχρεωτικό το σύστημα αυτό. Αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε στόχο μα ε, είναι να βρούμε αποτελέσματα. Αν όχι αυτό, να βρούμε κάποιο άλλο τύπο ρύθμιση. Πολλοί μίλησαν για περιφερειοποίηση. Ο κύριος Κάλαχερ, η κυρία Λεβίν και άλλοι Νομίζω ότι σχεδόν όλοι το ανέφεραν αυτό κάποια στιγμή. Να σας πω ότι είναι λίγο θολό το τι εννοούμε όταν μιλάμε για περιφερειοποίηση. Εγώ πιστεύω ότι σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι έχουμε διάφορα οικοσυστήματα, διάφορες ε, παραδόσεις, διάφορου τρόπου αλλίε. Χρειαζόμαστε όμως κοινή ρύθμιση, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να πετύχουμε διαφάνεια και περιφερειοποίηση. Αν μπορούμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να το συζητήσουμε. Θα πρέπει όμως να ε, διασφαλίσουμε τις σωστές επιθεωρήσεις, ε, επίσης ε, τη βιωσιμότητα του συστήματος, τη διαφάνεια, την δημοκρατικότητα του συστήματος. Αυτά νομίζω ότι είναι σημαντικά όταν μιλάμε για περιφερειοποίηση. Εάν είναι δυνατόν να το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις σας να πω ότι είναι σημαντικό όταν κοιτάμε το μέλλον ε, να βρούμε τρόπους ε, ρύθμισης και διαχείρισης των κοινών αλλιευμάτων μας που να μην ε, αφήνουν περιθώριο για απορρίψεις, να μην έχουμε διαμάχες ανάμεσα στους επιθεωρητές και τους αλληλείς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην οδηγηθούμε σε ε, αγώνες, σε μάχες ανάμεσα στους επιθεωρητές και τους αλληλείς. Να ενθαρρύνουμε τους αλληλείς να είναι υπεύθυνοι. Όχι να πολεμούν τους ε, επιθεωρητές. Νομίζω ότι αυτός είναι καλός τρόπος να προχωρήσουμε και χρειαζόμαστε έναν τέτοιον κανονισμό για να έχουμε ε, αυτή την πρόπτικη. Τότε θα έχουμε βιωσιμότητα την οποία χρειαζόμαστε. Τότε θα μιλάμε για αλληλεία για το μέλλον. Και κάποιος αναφέρθηκε στην υδατοκαλλιέργεια. Χρειαζόμαστε περισσότερα ψάρια, χρειαζόμαστε βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες. Χρειάζεται να μπορούμε να ταΐσουμε όλους τους ανθρώπους με υγιεινά ψάρια, τα οποία μπορούμε να καλλιεργήσουμε στο μέλλον. Ας το κάνουμε αυτό λοιπόν. Η Προεδρία μου διαρκεί έξι μήνες. Η Ευρώπη εργάζεται και είμαι ανοιχτή ανα πάσα στιγμή ε, σε διάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Πέντε έχουν ζητήσει ακόμα το λόγο. Ένα λεπτό καθένας. Ο κύριος Ντέιβις πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, όσον αφορά τη δικασία, όσον αφορά τη διαδικασία. Δεν θα πετύχετε κοινή θέση μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Τι περιμένετε όμως ότι θα πετύχετε ως Προεδρία μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Όσον αφορά τα TFCs, είπατε ότι η Δανία πιστεύει ότι πρέπει να προχωρήσουμε με την πρόταση αυτή εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να απαγορεύσουμε τις παραχωρήσεις αυτές, τουλάχιστον να δώσουμε ευελιξία στα κράτη-μέλη, να δώσουμε ένα περιθώριο ευελιξία στα κράτη-μέλη, προκειμένου να σχεδιάσουν τα προγράμματα τα δικά τους. Καταλαβαίνετε ότι ε, η πιο εύκολη λύση βέβαια θα ήταν να επιβάλλουμε υποχρεωτικά το σύστημα αυτό στα κράτη-μέλη. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να δούμε πώς τα κράτη-μέλη θα καταφέρουν να μειώσουν την υπερβολική ικανότητα την ελευτική. Ο κύριος Ρωμέβα. Ευχαριστώ. Κάποια σχόλια, κάποια θέματα που ήθελα να θίξω ήδη έγιναν ε, για την περιφερειοποίηση συγκεκριμένα. Ε, λείπει μία έννοια, η συνδιαχείριση, co-management. Πώς την πρόταση αυτή μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κάποια τμήματα του τομέα, κυρίως ε, όσοι λειτουργούν υπεύθυνα ε, και μιλώ και για τον αριστικό ε, στο τεχνικό τμήμα του κλάδου, πώς μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία. Και δεύτερον, χτες στην Επιτροπή δύο φορές ψηφίσαμε την αναγκαιότητα ε, να καταρτιστούν ε, σχέδια ε, μακροπρόθεσμα για την ανασύσταση του πληθυσμού πάνω από το MSY, τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Αυτή θα είναι μία από τις μάχες που επίσης θα δώσετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ευχαριστώ, η κυρία Πατράου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Υπουργό που περιβρίσκεται εδώ, τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις. Καταρχήν, για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Μεγάλες προσδοκίες ε, στην αρχή, στη συνέχεια σταμάτησε κατά κάποιο τρόπο ε, και είναι πολύ σύντομο το χρονοδιάγραμμα. Ποιο είναι το επίπεδο της δέσμευσης της ε, Προεδρίας της Δανίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Δεύτερον, μιλήσατε πολύ για την αηφορία Πρέπει να επαναλάβω. Καταλάβατε τι είπα. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Αηφορία. Μιλήσατε πολύ για την αηφορία. Η Επίτροπος τελευταία άρχισε να μιλάει για μια καθολική αηφορία που θα περιλαμβάνει την κοινωνική πτυχή, την οικονομία και το περιβάλλον. Άκουσα να αναφέρεται τα ε, περιβάλλον και την οικονομία, αλλά δεν άκουσα το κοινωνικό κομμάτι και Τρίτο θέμα, εξωτερική διάσταση. Πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αποτελεί το παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο με μέτρα αρκετά πιο περιοριστικά. Με ανησυχεί αυτά τα περιοριστικά μέτρα πολλές φορές ε, θίγουν τον ελευτικό τομέα. Ναι, να έχουμε περιβαλλοντική εφορία, αλλά μέσα σε ένα καθολικό πλαίσιο. Ευχαριστώ την κυρία Πατράου. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Προεδρία για τη δυνατότητα που μας δίνεται για την ανταλλαγή απόψεων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποκέντρωση είπατε ότι είναι ασαφή και συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ όμω ότι χρειαζόμαστε κοινού κανονισμούς, κοινή ρύθμιση, κοινού στόχους χρειαζόμαστε και θα επωφεληθούμε πολύ περισσότερο αν αποκεντρώσουμε τελικά την, το μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Δεν χρειαζόμαστε ρυθμίσεις και κανονισμούς σαν αυτούς που έχουμε τώρα στα πλαίσια της κοινή ελευθερικής πολιτικής όσον αφορά τις απορρίψεις. Δεν χρειαζόμαστε τους κοινού αυτούς κανόνες. Χρειαζόμαστε συνεργασία κοινούς στόχους και θα καταφέρουμε να καταλήξουμε τελικά σε ρυθμίσεις πολύ πιο αποτελεσματικές όσον αφορά τις μεταβάσιμες ελευτικές παραχωρήσεις. Η Δανία κατέδειξε ότι δεν χρειάζεται να έχουμε κοινέ υποχρεωτικές απαιτήσεις για τα TFCs. Εθελοντικά και εφόσον κρίνεται ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ωφελήσει τα κράτη-μέλη, τότε μπορούν να το κάνουν. Διαφορετικά, δεν είναι δυνατόν να έχουμε όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τα TFCs και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα οδηγούσε και σε διεθνείς τέτοιες μεταφορές παραχωρήσεων και με κατάφου του πράγματος. Ο κύριος ε, Σάντσες, ε, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Υπουργό για την ε, παρέμβασή τη και θέλω να ευχηθώ και κάθε επιτυχία στην ε, Δανική Προεδρία. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια τη Προεδρία σα πρέπει να προσδώσετε μεγαλύτερη αξία στον ε, κλάδο και να σα πω ότι το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτη και πρέπει να ελέγχει την εφαρμογή τη νομοθεσία σα. Και καθώ υπάρχει αλλαγή του ρόλου του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να προωθηθεί. Επίση, η κοινωνική διάσταση είναι σημαντική γιατί ο κλάδος είναι πρωταγωνιστής στην μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προστατευτεί ε, και είναι απαραίτητο να είναι αποτελεσματική μεταρρύθμιση, όχι να μείνει μόνο στα χαρτιά. Και τρίτο, για το Μαρόκο έχουμε μία λευτική συμφωνία, λείπει το πρωτόκολλο και απορρίφθηκε η παράταση του πρωτοκόλλου, αλλά ταυτόχρονα ζήτησε το Κοινοβούλιο και νέο πρωτόκολλο. Εγώ θέλω να σας ζητήσω να μην ε, πληρώσει ο λευτικός ε, τομέας ε, την σχέση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Μαρόκο και θεωρούμε ότι τα προβλήματα που έχουμε και σε άλλους τομείς πρέπει να αντιμετωπιστούν και να λυθούν με την ίδια, να υιοθετηθεί η ίδια λύση. Ε, η κυρία Γκαρσία, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Υπουργό τηλεγραφικά να σας πω ότι συμφωνώ με τα ουσιαστικά θέματα που έθιξαν οι δύο συνάδελφοι, η κυρία Φράκα όπως ε, ε, και ο κύριος Σάντσες. Ε, δεν θα αναφερθώ λοιπόν στα σχόλιά τους αλλά θα αναφερθώ στο πρωτόκολλο που δεν κυρώθηκε στο πρωτόκολλο της συμφωνίας με το Μαρόκο. Δεν ξέρω να έχετε σκεφτεί τις συνέπειες που επέφερε αυτό και ποιες συνέπειες θα μπορούσε να έχει στο μέλλον, δηλαδή να μην ε, υπογραφεί το νέο πρωτόκολλο, γιατί όλοι με τα λόγια μπορεί να αισθανόμαστε πολύ άνετα, αλλά θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο λαός της Δικής Σαχάρας ε, δεν ε, παραβίαζονταν τα δικαιώματά του δυνάμει τη της συμφωνίας, αλλά ωφελούνται από τη συμφωνία αυτή. Ο κίνδυνος είναι όσοι ελεύουν τώρα 90% που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε ε, τις ε, τεχνικές ε, για την περιβαλλοντική εφορία μπορούν να το κάνουν και αν ε, εμείς ε, που έχουμε την ευθύνη για την κυβέρνηση για να διαφυλάξουμε τα κοινωνικά, τα περιφελοντικά συμφέροντα και τα συμφέροντα των πολιτών ε, δεν δράσουμε τότε θα έχουμε πολύ αρνητικές συνέπειες. Έτσι λοιπόν θέλω να ζητήσω το νωρίτερο να εκπονηθεί ένα νέο πρωτόκολλο. Μάλιστα, κύριε Υπουργό, για να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σα και για το χρόνο σα. Έχετε το λόγο. Φυσικό θα μείνω, διότι νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τη δυνατότητα ε, αυτού του ε, άμεσου διαλόγου μαζί σας ε, για διάφορα θέματα. Διάφορες ερωτήσεις τέθηκαν. Κύριε Ντέιβις, ρωτήσατε ποιες είναι οι προσδοκίες μας όσον αφορά την γενική προσέγγιση τον Ιούνιο. Συμφωνώ μαζί σας. ότι θα ήταν προτιμότερο αν έχουμε προαιρετικές ε, μεταβάσιμα αληφτικές παραχωρήσεις, ε, να ε, συζητήσουμε το θέμα της αληφτικής ικανότητας. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το scrapping. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση, αλλά θα μπορούσε να είναι μια συζήτηση, αλλά μόνο εφόσον δεν δεχτούμε νέα σκάφη αυτά για το scrapping, τον παροπλισμό. Ε, αρκετοί από εσά αναφέρθηκαν στα μακροπρόθεσμα προγράμματα διαχείρισης. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι ε, αυτό το πρόγραμμα αποτελεί αντικείμενο ε, συναπόφασης όσον αφορά κάποια είδη, όσον αφορά το σαβρίδι, ε, υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Εμείς ως Προεδρία προσπαθούμε να βρούμε λύση, ε, να βρούμε κοινό τόπο, να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις με ανοιχτό μυαλό και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει, διότι δύο μέρη έχουν οι διαπραγματεύσεις αυτές και εμείς από την πλευρά μας είμαστε πολύ ανοιχτοί. Όσον αφορά το Μαρόκο, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό. Ακούω φωνές από χώρες όπου το θέμα αυτό είναι σημαντικό οικονομικό θέμα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε εποχές οικονομικής κρίσης. Επίσης όμως πιστεύω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι εσείς, εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο, σταματήσατε το πρωτόκολλο, το ενδιάμεσο πρωτόκολλο. Το σημειώνουμε αυτό στο Συμβούλιο. Μη μου πείτε ότι δεν έχει σημασία αυτό που κάνετε, διότι εδώ ε, είχατε πολύ σημαντική επιρροή στο θέμα αυτό. Αυτό σήμαινε, σήμανε ότι ε, τώρα διαπραγματευόμαστε νέα διαπραγματευτική εντολή για την Κομισιόν. Με τη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή είναι πιο σφιχτή διαπραγματευτική εντολή. Προσεγγίζει και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βιωσιμότητας. Ε, μιλάμε για αλία πλεονασμάτων. να δοθούν ευκαιρίες στο, στο λαό της Δυτικής Σαχάρας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή εντολή αυτή, συζητιέται στις ε, ομάδες εργασίας και νομίζω ότι γρήγορα θα προχωρήσει. Μετά όμως θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο και μετά θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Παρότι λοιπόν προσπαθούμε να εργαστούμε γρήγορα, είναι μια μακρόχρονη διαδικασία θα διαρκέσει κάποιο χρόνο. Έτσι ε, αντιλαμβάνομαι τη δουλειά που γίνεται στην Κομισιόν και στις ομάδες εργασίες. Όσον αφορά την βιωσιμότητα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι η βιωσιμότητα αφορά κυρίως το περιβάλλον. Είναι όμως επίσης σημαντικό ε, να είναι και οικονομικά βιώσιμο ό,τι κάνουμε. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι δυνατό να έχουμε παράκτια αλληλεία και στη νέα με αυτή μεταρρύθμιση. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε και την διαχείριση των ε, αλληλευτικών αποθεμάτων μας. Θα πρέπει όλοι να προχωρήσουμε λοιπόν με ανοιχτό μυαλό στις διαπραγματεύσεις αυτές. Υπόθηκε ότι δεν χρειαζόμαστε κοινό στόχο, δεν χρειαζόμαστε κοινή νομοθετική ρύθμιση, χρειαζόμαστε κοινού στόχους. Συμφωνώ με την έννοια ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι, με αυτήν, την, ότι σε αυτήν τη μεταρρύθμιση είμαστε 27 χώρες. Δεν είμαστε πια 17, 15, είμαστε 27 χώρες. Και αυτό επηρεάζει τον τρόπο που ρυθμίζουμε την νομοθεσία και θα πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια μεταρρύθμιση που να μας δώσει βιωσιμότητα, νέες θέσεις απασχόλησης, ανάπτυξη, ε, που θα μας δώσει επίσης υγιεινά τρόφιμα, λιγότερη γραφειοκρατία περισσότερη ευθύνη για τους αλληλείς και διαφάνεια για όλους μας. και για μας που νομοθετούμε και για τους επιθεωρητές. Αυτό θέλουμε, ας το συζητήσουμε. Επί έξι μήνες θα βρίσκομαι εδώ ως πρόεδρος του Συμβουλίου. Ε, Ξεκινήσαμε σήμερα τον διάλογο. Ε, ας υποσχεθούμε όμω ο ένα τον άλλον να μην τον σταματήσουμε σήμερα, να συνεχίσουμε το διάλογο αυτό κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και ελπίζω ότι ε, οι προσδοκίες που θέσαμε στην ε, Προεδρία σας, που έχουμε από την Προεδρία σας, ε, να καταστούν πραγματικότητα το επόμενο εξάμεινο. Θα χαιρετήσουμε τον κύριο Υπουργό και θα συνεχίσουμε σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πριν ε, να ξεκινήσουμε το σημείο 14, κυρία Φράγκα. Ναι, θα ήθελα να πω κάτι. Και δεν θα μπω τώρα σε επίμαχα ζητήματα, αλλά θέλω να θίξω ένα θεσμικό ζήτημα. Η κυρία Υπουργό είπε ότι τελικά για τα θέματα συναπόφαση όπω τα σχέδια διαχείριση. Αυτό είναι ε, κάτι που πρέπει να ρυθμιστεί μεταξύ των δύο μερών και να έχουν και οι δύο καλή θέληση. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτοί που έχουν δείξει την καλή θέληση εδώ ήταν μόνο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχε συνέχεια όλο ένα και πιο περιοριστικές θέσεις και δεν είχε ποτέ την πρόθεση να συνάψει συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα αυτό να είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα θα το γράψω στα πρακτικά. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δυστυχώς ε, δεν γνωρίζω την κατάσταση αυτή. Πάντω πιστεύω ότι οποιοδήποτε μέλος αυτής της ε, Επιτροπής ε, μπορεί πάντοτε να ζητά το λόγο και φυσικά υπάρχει απόλυτη ναι. ευελιξία σε αυτό ακόμη ε, και αν πρόκειται και παρουσία της εκπροσώπου της Προεδρία, Προεδρίας θα πρέπει να παίρνουν το λόγο βουλευτές γιατί έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Λοιπόν, ε, σημείο 14, μεταρρυθμίσει κίνηση ελευτική πολιτική. Για δεύτερη φορά θα δούμε αυτό το θέμα. Και χωρί χρονοτριβή, να δώσω το λόγο στον κύριο Σελαβράκο για να μα παρουσιάσει τι εργασίε του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, ξέρετε καλύτερα από μένα όλοι ότι η Αλία, όπως όλη η ανθρωπότητα και όλη η οικονομία, βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής σε αυτό το σημείο καλούμεθα να κάνουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις αφού κατά κοινή ομολογία η κοινή αλλιευτική πολιτική που προηγούμενα είχε καθιερωθεί παρουσιάζει ορισμένα κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Ε, είναι ανάγκη λοιπόν να κάνουμε την αλληλεία προσαρμοσμένη στο περιβάλλον, περιβαλλοντολογικά λοιπόν, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμη. Η Ένωση και τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν στις παγκόσμιες διασκέψεις του Ιωάννησμου και της Ναγκόγια για να δράσουν κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών ηχθιαλιβάτων και ηχθιαποθεμάτων με σκοπό την αποκατάσταση των επιπέδων εκμετάλλευσης ε, των εμβίων πόρων σε επίπεδα ικανά να παράγουν μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή προτείνει στο βασικό κανονισμό να καθοριστεί για κάθε είδος η μέγιστη βιώσιμη απόδοση η οποία ορίζεται ως η μεγαλύτερη ποσότητα λιευμάτων που μπορεί να λαμβάνεται με ασφάλεια για αόριστο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή, από ό,τι διάβασα, ορίζει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2015 για την επίτευξη της MBA. Ε, η επίτευξη του στόχου παραγωγής μεγίστης βιώσης απόδοσης για όλα τα αποθέματα μέχρι το 2015 είναι ευκταία βέβαια αλλά στην πράξη φοβούμε ότι δεν είναι βιολογικά εφικτή. Η προσέγγιση της Επιτροπής ίσως πρέπει να αναθεωρηθεί δεδομένου ότι γίνεται λόγος για όλα τα αποθέματα ακόμη και αν προέρχονται από μεικτή ελία. Το θέμα θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω και να δοθούν απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων που προκύπτουν ως προς την επιστημονική βάση στην οποία στηρίζεται η πρόταση και τη δυνατότητα επίτευξη του στόχου ανά όπου είναι εφικτό για το 2015 και για τα υπόλοιπα μέχρι το 2020 προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι ίσως είναι πιο σωστό και ρεαλιστικό να διατηρήσουμε τη διατύπωση που υιοθετήθηκε στην παγκόσμια διάσκεψη του Γιωχανέσμου ε, διατηρώντας τον ορισμό του MBA τον όρο όπου είναι δυνατόν. Ε, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να έχω τις απόψεις των συναδέλφων και των σχεδόν εισηγητών πάνω σε αυτό το θέμα καθώς και, το, και τις απόψεις της Επιτροπής διότι ε, πιστεύω ότι η προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε πρέπει να είναι περισσότερο συλλογική διότι θα έχει αποτελέσματα και επιπτώσεις πάνω στην κοινή αλλιευτική πολιτική της Ένωσης για πολλά χρόνια. Και βλέπω και χαίρομαι ιδιαίτερα που οι συνάδελφοι στην Επιτροπή αυτή είναι εξειδικευμένοι τόσο καλά που τους θαυμάζω ειλικρινώς. Ε, κρίνω σημαντική τη συμμετοχή των αλλιέων και των φορέων του κλάδου για τη συλλογή ασφαλών συμπερασμάτων και ίσως ε, θα πρέπει ε, να δούμε και επιτροπές αλλιέων και επιτροπές αρμοδίων πάνω στο θέμα της αλίας για να βγάλουμε σαφή συμπεράσματα. Η αξιοπιστία των επιστημονικών δεδομένων. Μια πολιτική τέτοιου είδου δίδει προφανώ προτεραιότητα στην αξιοπιστία των επιστημονικών δεδομένων και η διαθεσιμότητά τη πρέπει να τεθεί ω μία από τι σημαντικότερε προτεραιότητε τη μεταρρύθμιση αυτή. Σε ορισμένε γεωγραφικέ περιοχέ, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, πέρα από την έλλειψη δεδομένων, η σημαντική παρουσία τη μεικτή αλληλεία καθώς και η επαλληλία των εθνών ζωνών αλληλίας καθιστά δύσκολη τη συλλογή δεδομένων για την αποτελεσματική εφαρμογή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα στην προκειμένη περίπτωση. Η συλλογή των δεδομένων είτε ως μέσο είτε ως στόχος παρόλο που απαιτείται ως προϋπόθεση για τη λήψη μέτρων διαχείρισης των αποθεμάτων θεωρώ ότι θα πρέπει να προϋποθέτει την τήρηση των ίδιων διεθνών κανόνων και την κύρωση διεθνών συμβάσεων και ειδικότερα την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας με τα συνεργαζόμενα μέρη. Για να είναι αποτελεσματική η κοινή αλλιευτική πολιτική, ίσως είναι απαραίτητο να στηρίζεται σε ποιοτικά επιστημονικά δεδομένα και να συντονίζει τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων κάθε κράτους μέλους. Στην ανακοίνωσή της, αναφέρεται ότι η Επιτροπή μελετά ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα για τη διαχείριση της αλληλείας. Κάτι τέτοιο κρίνεται πολύ σημαντικό για τον συντονισμό και την παραγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Η εκπόνηση εθνικών προγραμμάτων έρευνα θα πρέπει να τύχει τη οικονομική υποστηρίξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τούτο θα προκύψει από το άτομο 38 του κανονισμού. Ε, η πρακτική της εξάλληψης των απορρίψεων η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρακτική μέχρι το 2016 είναι εφικτή και προτείνει την εξάλληψή της. Θεωρώντας δικαίως ότι οι απορρίψεις καταρχήν είναι απαράδεκτες. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Οι απορρίψεις είναι απαράδεκτες. Λόγω κυρίω της διμενούς επίπτωση σε σειρά αξιολογήσεων ζωτικής σημασίας. Δεν ξέρω πόσο ε, ε, τούτο ε, είναι εφικτό. Συγγνώμη. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη διερμηνία στα αγγλικά. Λύθηκε, ωραία. Uh, I'm going very, very Okay? Υπάρχει κάποιος θόρυβος και όχι διερμηνία, λέει ο πρόεδρος. De acuerdo, adelante. Προχωρήστε, eh, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι ο Όσκορ Βάιλντ είχε πει ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για την πρώτη εντύπωση. Εγώ αυτή τη στιγμή <laughs> είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω και λόγω του προβλήματο παρακαλώ να μου δώσετε δεύτερη ευκαιρία. Ε, επανέρχομαι. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξάλληψη των απορρίψεων μέχρι το 2016 είναι εφικτή. Ε, μακάρι στην πράξη αυτό να ε, φανεί ότι είναι ικανοποιητικό και μπορεί να επιτευχθεί. Φοβούμε όμως ότι ίσως είναι εκτός ε, κοινή λογικής και θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο. Το θέμα είναι σύνθετο, ιδιαίτερα στο επίπεδο της πολυειδικής αλληλείας και είναι αναγκαίο να αναλυθούν καταρχάς οι λόγοι που οδηγούν στις απορρίψεις ώστε να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία αναπερίπτωση όπως η βελτίωση της επιλεκτικότητας των εργαλείων αλλίευση και αθώς και η εκπαίδευση και η ενημέρωση των αλλιέων. Ξέρετε ότι ε, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο που έχω μια εμπειρία η αλληλεία μεταβάζεται από πατέρα σε γιο χωρίς ειδικότερη εκπαίδευση και ενημέρωση και δεν παρουσιάζεται στους νέους αλληλείς η εκπαίδευση εκείνη που χρειάζονται με τα νέα δεδομένα να ασκήσουν την αλληλεία. Και έχουμε πρόβλημα. Συμφωνώ επίσης με τη βασική αρχή της μείωσης των απορρίψεων. Θεωρώ όμως ότι η εξάλληψη δεν θα είναι ρεαλιστική. Το μέτρο κατά την άποψή μου πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον σύστημα ποσοστώσεων και να προσδιοριστούν οι μηχανισμοί υπολογισμού των απορρίψεων, να συνεκτιμηθεί το διοικητικό κόστος και οι δυσκολίες της επιθεωρήσης της ελίας, το πώς ελέγχεται. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρώ θετική την ιδέα να αναπτυχθεί ένα πιλωτικό σχέδιο ή πιλωτικά σχέδια προκειμένου να διαπιστωθούν οι τεχνικές δυσκολίες και το κοινωνικό και οικονομικό κόστος του μέτρου αυτού πριν από τη γενίκευση της εφαρμογής του. Θα ήταν καλό να γίνουν περαιτέρω μελέτες και να ληφθούν υπόψη οι διάφορες αλληλευτικές τεχνικές, κατά την απόψη. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη σημασία της ψυχολογίας του κλάδου για τη εταιρική ανάλυση, από αυτό εξαρτάται και η αποτελεσματική εφαρμογή ενός μέτρου. Η υποχρέωση διάθεσης κάποιων αλλιευμάτων για ηχθιάλευρα ή ζωοτροφές προϋποθέτουν την ύπαρξη σχετικών εγκαταστάσεων. Αντιλαμβάνεστε, όπως είναι δομημένες οι διάφορες γεωγραφικές περιοχές, έχουν και τις ιδιαίτερες συνθήκες τους, όπως είναι η Μεσόγειος, αλληλεία μικρής κλίμακος, πολλά μικρά απομονωμένα νησιά και μικρά λιμάνια, δύσκολες υγειονομικές συνθήκες λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να μιλάμε τα ίδια μέτρα για την Βαλτική, για τη Μεσόγειο, για τον Πόνο. Λείπει από την πρόταση της ε, Επιτροπής από τη μια συνολική προσέγγιση ε, με την οποία θα πρέπει αυτά τα σχέδια να περιλαμβάνουν ε, μια πλήρη αντιμετώπιση του θαλασσίου περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος για να μπορέσουν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη μείωση της παραλίευσης των πόρων πρέπει να βάλουμε και την οικολογία στη ζωή μας, δεν είμαι οικολόγος, αλλά θεωρώ πλέον ότι οι ανάγκες όπως εξελίσσονται καθιστούν την οικολογία ένα σημαντικό κομμάτι των προβληματισμών μας σε οποιαδήποτε κοινωνική και οικονομική μας δραστηριότητα. Οι αλληλείς θα πρέπει να έχουν ένα κεντρικό ρόλο στη συνδιαχείριση και τον σχεδιασμό αυτών των αποθεμάτων και αν αυτό καταστεί εφικτό θεωρώ ότι ίσως ε, θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Το σύστημα των ατομικών μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων, το TFC. Ο προτινόμενος βασικός κανονισμός καθιερώνει ένα βασιζόμενο στην αγορά κίνητρο για τη δημιουργία ενός ισχυρού κερδοφόρου αλληλευτικού κλάδου μέσω της σταδιακής εφαρμογής των μεταβιβάσιμων αλληλευτικών παραχωρήσεων θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της εμπαραγματοποίησης του δικαιώματος πρόσβασης στους πόρους και του γεγονότος ότι οι αλληλευτικοί πόροι αποτελούν δημόσιο αγαθό. Επίσης, θα πρέπει να προευθούν ρήτρε διασφάλισης και ικανά εχέγγυα για να προστατεύσουν την αλληλεία μικρής κλίμακος και την παράκτη αλληλεία για να, να μην δημιουργηθούν οικονομικές και κοινωνικές ανισορροπίες. Η περιφερειοποίηση είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο δεν πρέπει να παραμείνει στο wishful thinking αλλά πρέπει να γίνει πράξη. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει ε, να ενώσει και την Ευρώπη περισσότερο. Η αναφορά νομικής βάσης απαιτείται καθώς και περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο υιοθέτηση και εφαρμογής είναι άμεσα ενδιαφέρουσες. Η Επιτροπή προτείνει περιφερειακά μοντέλα συνεργασία και ειδικότερα στην περίπτωση του ευξήνου πόντου την δημιουργία γνωμοδοτικού συμβουλίου ευξήνου πόντου για την ανταλλαγή απόψεων με τέσσερα κράτη-μέλη που δεν είναι και μέλη της Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για τη Μεσόγειο. Η διασαφήνιση του πλαισίου καθίσταται επιτακτική και όπου η υιοθέτηση του συστήματος ενδέχεται να περιλάβει και τρίτες χώρες διότι ε, ξέρετε ότι έχουμε και ω προς το υπογάστριο το ευρωπαϊκό της Αφρικής, κοινά θαλάσσια σύνορα. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και της Επιτροπής και των αποφάσεων και των ε, δικών μας ε, προβληματισμών με διαφορετικές πολιτικές για να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν καλύτερες πρακτικές η ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας και οι αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες εν ώψη της μεταρρύθμισης τέτοιας κλίμακος πρέπει να προβλεφθούν και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην διατήρηση επαγγελματιών ψαράδων οι οποίοι θα κάνουν ένα ψάρεμα το οποίο δεν θα παραβιάζει το περιβάλλον και θα έχει και τη μέγιστη απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό συνάμα πρέπει να δούμε την αύξηση του τομέα υδατοκαλλιέργειας, το οποίο μπορεί να προσφέρει καλή και συνεχή απασχόληση. Ε, όλα αυτά τα οποία λέγω πρέπει να συνδυαστούν ε, με την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ένωση, διότι για όλα όσα λέμε χρειάζονται χρήματα. Ε, θέλω να πιστεύω ότι λαμβανομένου υπόψη ότι σαν οικονομικού παράγοντος στη διαμόρφωση του εισοδήματος των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ελία έχει μεγάλο και σημαντικό μέρος. Θα βρούμε τα κατάλληλα χρήματα ή τουλάχιστον θα ξεκινήσουμε καλά. Ε, θα παρακαλούσα πάρα πολύ στο σημείο αυτό για τη βοήθεια όλων σας στο να γίνει κάτι καλύτερο σε αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Σελαβράκο. Καταρχήν ο κύριο και η κυρία Λέβετ στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την έκθεση αυτή, πολύ χρήσιμη. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη μπορώ να υποβάλω τροπολογίες για την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την Κοινή Αλληλευτική Πολιτική θα χρησιμοποιήσω το έγγραφο αυτό λοιπόν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για να προσπαθήσω να ε, τροποποιήσω κάποιε από τι ε, ιδέες που θέλω να, ε, ε, υποβάλω. Κάποιε παρατηρήσει. Ο ορισμό για το σκάφο αλληλεία σε μικρής κλίμακα. Συνήθως είναι μικρότερο από 10 μέτρα, 12 μέτρα στην πρόταση για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Αναφέρθηκε ότι στην Ιρλανδία στην Ιρλανδία είναι μεγαλύτερα τα μικρά σκάφη. Φαντάζομαι γιατί θα μπορούσε κανείς να θέλει να χρησιμοποιήσει κάπως μεγαλύτερα σκάφη. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το λύσουμε αυτό. Για τις πρώτες σας ερωτήσεις, ε, το 2015 ως ε, ε, έτος αναφοράς για το MSY για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ξέρουμε ότι το 2015 δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να προλάβουμε την προθεσμία αυτή, αλλά απ' την άλλη Θέλουμε νομική υποχρέωση. Ίσως θα πρέπει να ε, διατηρήσουμε το 2015 ε, και να πούμε ότι εντάξει δεν προλάβουμε όλες τις προθεσμίες, αλλά ε, αν δεν προλάβουμε τις προθεσμίες να προσπαθήσουμε να τα προλάβουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να, να το συμπεριλάβουμε αυτό στο, στην νομοθεσία και να δεχτούμε ότι δεν είναι εφικτό. Αν και βέβαια δεν είναι πολύ καλός τρόπος αυτός να νομοθετεί κανείς, αλλά μήπως είναι πρακτικός τρόπος. Δεύτερον, όσον αφορά την ισορροπία ανάμεσα στου ε, οικονομικού, κοινωνικού ε, και περιβαλλοντικού παράγοντε. Ε, φυσικά θέλουμε να πετύχουμε μια ισορροπία. Θέλουμε να φροντίσουμε να υπάρχει ο μέγιστο αριθμό θέσεων απασχόληση για του αλληλεί και θέλουμε επίση να διασφαλίσουμε την επιβίωση των παράκτιων κοινωνιών. Αλλά σε κανέναν άλλον τομέα, ούτε καν στη γεωργία δεν εξαρτιέται τόσο πολύ ο κόσμο επαγγελματικά από την φύση. Ο καλύτερο τρόπο λοιπόν να διασφαλίσουμε το μέλλον των ε, αλλιών είναι να αποφύγουμε την υπεραλίευση. Θα πρέπει ε, η οικολογία να είναι, απολύτως, ε, να είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Εάν δεν προσέξουμε την οικολογία δεν θα έχουμε καλό μέλλον για, την, για τον τομέα τη Το θέμα της επιστήμης, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχω δει έγγραφα εργασίας από την Κομισιόν που να εξηγεί πώς ε, θα ε, αντιμετωπίσουμε το κενό επιστημονικών στοιχείων. Ένα τεράστιο χάσμα αυτή τη στιγμή. Ε, μιλάμε για την αρχή της προφύλαξης στην περίπτωση όπου δεν έχουμε επιστημονικά στοιχεία, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι αρκεί, δεν είναι ικανοποιητικό. Ξέρω ότι τα κράτη-μέλη επί πολλά χρόνια είχαν την υποχρέωση να υποβάλουν τα επιστημονικά στοιχεία. Πολλοί στην Κομισιόν λένε ανεπίσημα ότι τα κράτη-μέλη αποφεύγουν να εκπληρώσουν αυτήν την υποχρέωσή τους, ε, απλά στέλνουν ε, τους ε, υπουργού απροετοίμαστου στις συναντήσεις του Δεκεμβρίου, ώστε να θέσουν την πολιτική πριν από την επιστήμη. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το θέμα... τις προθεσμίες του 2016 για την απαγόρευση των απορρίψεων. Είναι ρεαλιστική αυτή η προθεσμία. Το μεσημέρι πριν, ε, ένα μεσημέρι πριν τα Χριστούγεννα είχαμε μια παρουσίαση από τον ε, πρώην ε, Γενικό Διευθυντή της Αλλιές της Νορβηγίας που ήταν ε, ε, αρμόδιος τότε που η Νορβηγία ε, εισήγαγε την απαγόρευση απόρριψης κατά τη δεκαετία του 90. Είχε πει τότε στον Υπουργό του ότι θέλουμε να μειώσουμε τις απορρίψεις. Δεν είναι πρακτικό αυτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε τόσο γρήγορα. Ο Υπουργός επέμενε, είπε ότι όχι, θέλω να γίνει αυτό, θέλω να γίνει κάντε το. Ε, και είχε δίκιο, διότι αυτό που έκανε ήταν ότι άλλαξε την οτροπία ε, στον ε, τομέα. ο κόσμος είχε αρχίσει να μιλάει για την εισαγωγή επιλεκτικών εργαλείων αλληλείας, αλλά με το που εφαρμόστηκε η απαγόρευση, το θέμα αυτό προωθήθηκε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι στην Νορβηγία ακόμα απορρίπτουν ψάρια οι αλληλείς, αλλά όχι τόσο πολύ, το κάνουν όταν δεν κοιτάει κανείς. έχουν μειωθεί πάρα πολύ όμως οι απορρίψεις, αποτελεί μέρος της λύση, παρότι δεν είναι ε, η, όλη η λύση. Θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση, διότι αυτή θα οδηγήσει σε καλύτερη πρακτική. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι σε αυτή την ε, άσκηση των προεδρικών κατευθυντικών συνεχώς θα συζητάω να μην μακρηγορείτε. Και το κάνω γιατί έχουμε χάσει πολύ χρόνο. Παρακαλώ κύριε Λέβιν και κατόπιν ο κύριο Κάντεκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σαλαβράκο για την έκθεσή σας ε, και το έγγραφο εργασία σας. Ε, περιέχει πολλά καλά στοιχεία και πολλά ε, πράγματα στα οποία συμφωνούμε και χαίρομαι πολύ που που βλέπω ότι τονίζεται και το καλό περιβάλλον που αποτελεί το μέλλον, τη βάση για το μέλλον οποιοδήποτε, οποιασδήποτε αλληλευτικής δραστηριότητας. Τονίζεται τα θέματα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης του MSY. Ε, αναφέρεται ε, αν είναι ρεαλιστικό ή όχι. Νομίζω το έχουμε συζητήσει αυτό στο παρελθόν με την Κομισιόν. Συμφωνώ με τον κύριο Ντέιβις ότι η μέγιστη βιώσιμη απόδοση μπορεί να αποτελέσει στόχο. Ξέρουμε ότι δεν θα τον πετύχουμε. Κάτι όμως που μπορούμε να πετύχουμε είναι Ε, η εκμετάλλευση των ε, αποθεμάτων ε, να γίνεται στα επίπεδα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση σε σχέση με τη βιομάζα. Δεν θα πρέπει λοιπόν απλά να πούμε ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η διατήρηση των αποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οικονομικά είναι καλύτερο, όπως έχει αποδειχθεί σε κάποια αλλιεύματα σε όλο τον κόσμο, αλλά τα αλληλευτικά αποθέματα θα πρέπει να διατηρούν ε, λειτουργία τους ως μέρος του οικοσυστήματος ε, που κρατάνε τους ωκεανούς σε ισορροπία. Τονίσατε τους ε, κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες επίσης. Είχαμε μια ακρόαση στο Κοινοβούλιο πριν τα Χριστούγεννα, δυστυχώς. Λίγο πολύ μόνο εγώ και η κυρία Φράγκα παρακολουθήσαμε αυτή την ακρόαση. Είχε να κάνει με την ανατροπή οικοσυστημάτων όταν η υπεραλίευση ε, αλλάζει ριζικά την τροφική αλυσίδα στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Είχαμε παρουσίαση μιας μελέτης με τίτλο «Η υπεραλίευση οδηγεί στα σε κιανοφίκη» και η απάντηση ήταν ναι. Η υπεραλίευση συμβάλλει σημαντικά ε, στο ε, καταστροφικό φαινόμενο των κοινοφικών και μάλιστα υπήρχε μία εκτίμηση στην έκθεση αυτή ε, σχετικά με τους... Ε, με το κοινωνικό-οικονομικό κόστος, μια συντηρητική εκτίμηση είναι 850.000 ευρώ το χρόνο. Στον υπολογισμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται καν όλα τα κράτη-μέλη. 850 εκατομμύρια, συγγνώμη. Ε, ε, υπάρχει λοιπόν πολύ σημαντικός κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος ε, εάν ε, είναι άρρωστη η θάλασσά μας. Αυτό επηρεάζει τον τουρισμό, την οικονομία και πολλούς άλλους τομείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα επίσης να πω ότι συμφωνώ απολύτως με το σημείο υπαριθμών 13 για τις απορρίψεις και τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μελλοντική μονοθετική ρύθμιση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσης να μην ενθαρρύνει τους αλλιείς να συνεχίσουν να αλλιεύουν τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα για να τα επικυρώσουν μετά. Θα πρέπει να ε, αποφεύγουν τα ε, παρεμπίπτοντα αλλιεύματα οι αλλοίς ε, και όχι να τα χρησιμοποιούν ως πρόσθετο ω πόρο πρόσθετου εισοδήματο. Και όσον αφορά την μικρή κλίμακα, νομίζω ότι τα 12 μέτρα είναι πολύ χοντρό εργαλείο, να το πω έτσι. Στην Σουηδία έχουμε ξύλινα σκάφη 20 ε, μέτρων που ε, αλλιεύουν με οικολογικό τρόπο, ε, αλλιεύουν μόνο κοντά στις ακτές και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτόν τον ορισμό. Αυτό λοιπόν είναι κάπως παράδοξο. Θα κλείσω εδώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Καντέκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Όσον αφορά τον ορισμό της αλίας μικρή κλίμακος, ο Κρις και η Ζαμπέλα μίλησαν γι' αυτό, σχετίζεται και με το ζήτημα τη περιφερειοποίησης πάντω ο ορισμό αυτό. γιατί η αλία μικρή κλίμακος δεν είναι ίδια στην Βόρεια Θάλασσα, στον Ατλαντικό, στη Μάνχη, στη Βαλτική Θάλασσα, διαφέρει από τη μία περιοχή στην άλλη. Επομένω το ότι δεν περιλαμβάνεται η έννοια της περιφερειοποίησης στην πρόταση μεταρρύθμισης κοινή ελευτικής πολιτικής δημιουργεί πρόβλημα ως προς τον ορισμό, ως προς την απόφαση για τον ορισμό της μικρής κλίμακος. Το είπε και η Ιζαμπέλα αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό και να ασχοληθούμε στα πλαίσια του βασικού κανονισμού. Όσον αφορά τώρα την μέγιστη βιώσιμη απόδοση, κύριε Σαλαβράκο, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εργασία σας. Σε κάθε περίπτωση ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι θα πρέπει να είναι ρεαλιστική η πρόταση όσον αφορά το έτος 2015, ιδίως όσον αφορά το ότι δεν έχουμε τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα ενδεχομένως ε, για κάποια είδη να καταφέρουμε να πετύχουμε την προθεσμία του 2013-2014, αλλά το να γίνει με τρόπο αποφασιστικό και καθοριστικό του 2015 θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο να οργανωθεί κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τώρα τις μηδενικές απορρίψεις, και στο σημείο αυτό συμφωνώ μαζί σας, Συμφωνώ με τις αμφιβολίες τις οποίες εκφράσατε όσον αφορά το ρεαλισμό μιας τέτοιας α, απόφασης. Καταλαβαίνουμε, ότι, όπως είπατε, ότι όλοι οι λιμένες δεν είναι το ίδιο εξοπλισμένοι και επομένως και υπάρχει και ένα ζήτημα ε, χαμηλού κέρδους ε, όσον αφορά τους ε, αλίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να καταφέρουμε να αυξήσουμε την δύναμη, την επιρροή που μπορούν να έχουν τα περιφερειακά συμβούλια, τα γνωμοδοτικά αυτά συμβούλια. Νομίζω ότι μπορούμε μέσα από τα συμβούλια αυτά να φτάσουμε στην επιθυμητή περιφερειοποίηση. Και κάτι ακόμα. Το να προασπίσουμε το περιβάλλον, τη διατήρηση των πόρων, προφανώς αυτό αποτελεί μία από τις ε, βασικές μας προτεραιότητες, έναν βασικό στόχο. Το να προασπίσουμε όμως αλύση είναι και αυτός ένας στόχος μας. Πιστεύω λοιπόν ότι οι δύο αυτοί στόχοι μπορούν να συνδυαστούν. Α σταματήσουμε λοιπόν να του φέρνουμε σε συνεχή αντίθεση και αντιπαράθεση. Γιατί από τη μια έχουμε αυτού που προασπίζουν ε, του πόρου και το περιβάλλον και από την άλλη αυτού που προασπίζουν ε, του αλληλεί. Θεωρώ ότι ο στόχο είναι κοινό. Αν δεν έχουμε πόρου, δεν έχουμε και αλληλεί. Είμαστε εδώ λοιπόν για να υπερασπίσουμε του αλληλεί, αλλά προφανώ και του φυσικού πόρου. Άλλο εξαρτώνται αυτά τα δύο. Ευχαριστώ, η κυρία Φράγα. Ευχαριστώ τον κύριο εισηγητή και θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Συμφωνώ ότι πρέπει να θέσουμε μία ημερομηνία. Εγώ θεωρώ ότι καλό είναι να θέσουμε το 2015, αλλά και με τις αποχρώσεις που έδωσε και ο κύριος Στίβενσον, δηλαδή να σεβαστούμε όσο αποφασιστήκαν στο Johannesburg στο μέτρο του δυνατού. Και κυρίως ε, γιατί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και επειδή θεωρώ ότι η πρόταση μεταρρύθμισης ε, της Επιτροπής εκεί η Κομισιόν προκαθορίζει ε, τις απορρίψεις και προκαθορίζει το θέμα της της βιώσιμης αποδόσης όμως εγώ νομίζω ότι τα σχέδια διαχείρισης είναι αυτά τα οποία συγκεκριμένα θα πρέπει να θέσουν αυτά τα στοιχεία ημερομηνίε, της βιώσιμη απόδοση απορρίψει κτλ. Γιατί δεν είναι το ίδιο να μιλάμε για απορρίψεις όταν ε, έχουμε ε, παραδείγματο χάρη αλλή ενός μόνο είδους όπου είναι λογικό να έχουμε πλήρη απαγόρευση των απορρίψεων το ίδιο δεν μπορεί να ισχύει για τις περιπτώσεις όπου έχουμε αλλία πολλαπλών ειδών μουλτισπίσης έτσι λοιπόν θα πρέπει πολύ συγκεκριμένα να καθορίζονται αυτά και αυτά θα πρέπει να καθορίζονται όπως είπα στα σχέδια διαχείρισης γιατί αυτό θα είναι το κυρίω στοιχείο της περιφερειοποίησης και εκεί πρέπει να δοθούν συγκεκριμένε αποχρώσεις και να συγκεκριμενοποιηθούν τα ζητήματα αυτά. Έτσι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι και το θέμα τη μέχρι τη βιώσιμη απόδοση αλλά και των απορρίψεων ε, και θα πρέπει να καθορίζονται συγκεκριμένα τα χρονοδιαγράμματα και ο τρόπος δράσης, όλα αυτά στα σχέδια διαχείρισης και έτσι θα υλοποιήσουμε τη περιφερειοποίηση. Σε ό,τι αφορά τώρα την παράκτη αιλία και τον ορισμό είναι ένα θέμα που συζητείται και μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο, αλλά όπως και να έχει και εγώ φοβάμαι πολύ ότι αν αυξηθεί το μέγεθος του σκάφους ε, της αεραστεχνικής αιλίας και τώρα που είναι στο να προστατεύουμε την αεραστεχνική αιλία ε, δεν θέλουμε να παρεκκλίνουμε από την πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι σωστά είναι τα όσα ανέφερε ο κύριος Σαλαβράκος. Εγώ συμφωνώ με το να υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση έτσι όπως τέθηκε, αλλά νομίζω ότι στα σχέδια διαχείρισης πρέπει να συγκεκρινοποιούνται όλα αυτά τα ζητήματα. Και όπως σας είπα, η Κομισιόν θέλει να προκαθορίσει τα πάντα. Επομένως, τι θα μείνει ε, να καθορίσει στα σχέδια διαχείρισης. Τελικά δεν θα έχουμε καμία περιφερειοποίηση. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, εμένα δεν μου αρέσει να μιλώ συνέχεια για το χρόνο, αλλά δύο, τρεις ακόμη βουλευτές ζητούν το λόγο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας δώσω το λόγο. Το αντίθετο, αλλά να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να περιορίσουμε το χρόνο των παρεμβάσεων ε, για να μιλούν και περισσότεροι και όχι να δίνουμε το λόγο σε λίγους μόνο, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Έτσι λοιπόν να δώσω το λόγο στους τέσσερις που τους ζήτησαν, αλλά σας παρακαλώ πολύ σύντομα και για τα επόμενα σημεία ναι, πρέπει να είμαστε πιο σύντομοι γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 12.30 και έχουμε ακόμα έξι σημεία. Ο κύριος Φερέιρα. Πρόεδρε, στην περίπτωση αυτή εγώ δεν θα μιλήσω γιατί εγώ θέλω διάφορα θέματα να θίξω και μπορώ να τα παρουσιάσω στην παρουσίαση της δικής μου έκθεσης. Μάλιστα, κύριε Πατράου. Μη Πρόεδρε, θα αναφερθώ μόνο στο θέμα του ορισμού της αριστεχνικής αλίας. Πολλές φορές ε, πρότεινα σε αυτό το βήμα να είμαστε κάπως πιο τολμηροί στον ορισμό αυτό και να μην περιοριζόμαστε μόνο στο μέγεθος του σκάφους. Αυτή είναι η ευκαιρία που έχουμε. Τώρα εμείς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα και μόνο ορισμό του small scale fisheries που θα καλύπτει όλη την επικράτεια. Χρειαζόμαστε έναν ορισμό πιο ευρύ, πιο ευέλικτο, που να περιλαμβάνει και περισσότερες ε, περιπτώσεις ε, και που ε, να μπορεί να καλύπτει κάθε γεωγραφική λεκάνη. Νομίζω ότι έχουμε αυτή την ευκαιρία και πρέπει να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε κυρία Πατράου. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά σωστά πράγματα υπόθηκαν ήδη και συμφωνούμε. Θα ήθελα όμως να αναφέρω ένα σημαντικό θέμα για μας στην Βαλτική και αλλού. Είναι η ε, σχετική σταθερότητα που, νομοθετη... που ρυθμίστηκε γύρω στο 1983 αλλά υπάρχουν συνεχείς διαμάχες μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις ποσοστάσεις κτλ. Εμείς θέλουμε σχετική σταθερότητα και ο αγαπητός συνάδελφος ε, Αλέν Καντέκ το ανέφερε και αυτό. Αυτό ήθελα να πω και όσον αφορά τις απορρίψεις. Πράγματι, πολύ σωστά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με τον ίδιο τρόπο που φτάσαμε μέχρι εδώ. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αποτελεσματικά τους πόρους μας. Ε, αν κάποιος έχει 10 ε, τόνους ε, σολομού και έχει έναν τόνο κάποιο άλλο ψαριού εκεί μέσα και, θέλει, και έχει εξαντλήσει την ποσόστοση για το σολομό, να απορρίψει το σολομό, όχι, αυτό είναι απαράδεκτο. δεν Θέλουμε να διατηρήσουμε την ε, αλία μας. Ε, αποτελεί μέρος της κληρονομιάς μας. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρο που μου δίνετε και εμένα το λόγο, πολύ σύντομα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για ένα πολύ χρήσιμο έγγραφο εργασίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει επικεντρωθεί στον ορισμό των μικρών αλλιευτικών σκαφών και της αλλίας μικρής κλίμακας. Κάποιος κάπου είπε ότι τα 12 ε, μέτρα θα πρέπει να αποτελούν το όριο. Αλλά συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν ε, ότι υπάρχουν ε, μεγαλύτερα σκάφη τα οποία είναι πολύ φιλικά προς το περιβάλλον. θα μπορούσαμε να έχουμε 15 μέτρα ως όριο, διότι τα σκάφη αυτά δεν είναι ούτε πολύ σύγχρονα, ούτε με πολύ εξειδικευμένο εξοπλισμό. Ε, αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κατανοώ ότι πολλά από τα θέματα που αναφέρθηκαν από τους κύριους βουλευτές είναι μεγίστο ενδιαφέροντος ε, και φυσικά αυτό είναι, ε, πολλά από αυτά θα τα συζητήσουμε λεπτομερώς γιατί έχουν να κάνουν με το βασικό κανονισμό αλλά θα ήθελα να τονίσω κυρίως θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο βασικό κοινωνισμό γιατί δεν είναι νομοθετικού χαρακτήρα, νομικού χαρακτήρα. Και νομίζω ότι αυτά είναι τα θέματα που είναι περισσότερο σχετικά στο πλαίσιο αυτής της γενικής ανακοίνωσης. Και θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της βελτίωσης των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Σίγουρα αυτό είναι ένας από τους μεγάλους στόχους ε, αυτής της μεταρρύθμισης, αλλά όπως σας είπα δεν είναι νομοθετικού χαρακτήρα, γι' αυτό δεν Βλέπετε συγκεκριμένες προτάσεις γι' αυτό στο βασικό κανονισμό. Πώς θέλουμε να το κάνουμε. Εκπονούμε ένα στρατηγικό έγγραφο το οποίο επικεντρώνεται σε τρεις μεγάλους τομείς, πώς θα καθορίζουμε τις προτεραιότητες για το μέλλον, πώς ε, θα αυξήσουμε τη χρηματοδότηση και το ανθρώπινο δυναμικό έτσι ώστε η επιστημονική κοινότητα στην Ευρώπη να μπορεί να απαντήσει σε προκλήσεις του μέλλοντος και πώς να βελτιώσουμε τη χρήση και ε, ε, των πόρων στην Ευρώπη, των επιστημονικών πόρων, γιατί υπάρχει ένας περιορισμός εκεί. πρέπει να συζητήσουμε το Μάρτιο σε μία συνεδρίαση ε, και με τους Γενικούς Διευθυντής Αλίας. Η Κομισιόν ε, προετοιμάζει ένα κείμενο προβληματισμού, ένα κείμενο συζήτησης για αυτή τη συνεδρίαση. Όταν αυτό το κείμενο προβληματισμού θα είναι έτοιμο, θα το στείλουμε στα κράτη-μέλη και παράλληλα ταυτόχρονα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν αποφασίσει αυτός ο οίκος ε, να κάνει μια συζήτηση με την Κομισιόν για το θέμα αυτό, φυσικά η Κομισιόν είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε. Και να προσθέσω κάτι ακόμα. Νομίζω ότι από τα διάφορα θέματα που ακούστηκαν, ε, νομίζω ότι ένα το ανέφεραν ε, όλοι οι παρεμβαίνοντες. Ε, ποιο είναι το κριτήριο για να ορίσουμε την αριστεχνική αλία ή την αλία μικρής κλίμακας. Νομίζω ότι εδώ στη θέση της Κομισιόν πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ ενός βασικού θέματος και ενός θέματος που το χρησιμοποιούμε εργαλείο. Δηλαδή το κύριο θέμα είναι ότι θέλουμε να έχουμε ειδικέ προϋποθέσεις για την μικρή κλίμακα σαλία. Πώς θα το ορίσουμε αυτό το κριτήριο των 12 μέτρων, ε, το έχω ξαναπεί. Φτάσαμε στο κριτήριο αυτό ουσιαστικά για τις που απαγωγή. Εξετάσαμε πολλά κριτήρια, κανένα από αυτά που εξετάσαμε δεν είναι τέλειο και θεωρούμε ότι αυτό των 12 μέτρων είναι απλό και είναι το λιγότερο ατελές, γιατί δεν εισάγει διακρίσει, είναι γενικό και επίση ε, στο πώς ε, μπορούμε να αξιολογήσουμε τους ε, στόλους ε, και πρέπει να έχουμε υπόψη και με τα 12 μέτρα. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό της ικανότητας και της ελευτικής ικανότητας στα πλαίσια της μικρής αριστεχνικής ελίας και σε όλα τα κράτη-μέλη ακόμη και αυτό το κριτήριο που σας φαίνεται πολύ περιοριστικό, αυτό που κάνει είναι το σε Ένα μεγάλο μέρο τη ε, θνησιμότητας ε, και του καθεστώτο που εφαρμόζεται για αυτή τη μικρή ελία αντιστοιχεί σε σκάφη 12 μέτρων. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν θεωρεί ότι τα 12 μέτρα δεν είναι το ουσιαστικό ζήτημα. Αν υπάρχουν ιδέε για το πώ να το βελτιώσουμε αυτό, βεβαίω ε, είμαστε ανοιχτοί να σα ακούσουμε. Όμως αυτό που τελικά χρειάζεται είναι ένα απλό και εύκολο κριτήριο. Μιλάμε πάντοτε για απλούστευση της πολιτικής μας. Αν τελικά έχουμε ένα κριτήριο που είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και δύσκολο να το ελέγξουμε και απαιτεί σημαντική προσπάθεια από τις εθνικές δικήσεις για να ελέγξουν αν κάποιος σέβεται ή δεν σέβεται τα κριτήρια για να εντάσσεται στον ορισμό του εραστέχνη ελιέα, τότε δεν απλουστεύουμε την πολιτική η Κομισιόν προσέχει πάρα πολύ το ζήτημα αυτό, αλλά ξέρετε θέλουμε και απλά κριτήρια και δίνουμε επίσης και ας δώσουμε επίσης ε, και πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της μη εισαγωγή διακρίσεων. Γιατί όταν ε, θα φτάσουμε στις διαθροτικές ενισχύσεις, ε, θα προτείνουμε διαθροτικές ενισχύσεις που για ένα σκάφος συγκεκριμένου μεγέθους ισχύουν σε μία χώρα και όχι σε μια άλλη. Προσοχή λοιπόν, γιατί μπορεί να προκύψουν διακρίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλαβράκος για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους οι οποίοι σχολίασαν την έκθεσή μου. Θεωρώ ότι είναι κοινή έκθεση όλων μας και προσπάθησα να συμπεριλάβω όλων τις απόψεις όπως έχουν ακουστεί και όπως έχουν διαμορφωθεί ε, στη διάρκεια της παρουσίας μου εδώ. Ε, θα συνεχίσω να είμαι σε επαφή, το γραφείο μου θα είναι σε επαφή με όλους τους συναδέλφους εις τρόπον ώστε μέχρι τη συντάξη του τελικού κειμένου να έχω τις απόψεις τους και τις παρατηρήσεις τους και αυτό θα αρχίσει από αύριο. Ε, εκείνο το οποίο θέλω να πω ως προς τα μήκη των σκαφών κατά την άποψή μου δεν είναι the main problem το μήκος του σκάφους. Διότι υπάρχουν οι ιδιαιτερότητες άλλο στις ανοιχτές θάλασσες, άλλο στην Μεσόγειο, άλλο στον Πόντο, στον Πόντο που είναι κλειστές οι θάλασσες και είναι διαφορετικές ε, οι δυνατότητες και οι ποσότητες των αλλιευμάτων. Εκείνο το οποίο είναι, είναι τα μέσα τα οποία θα πρέπει ίσως να μας προβληματίσουν τα, οποία, τα τεχνικά μέσα τα οποία ίσως ε, πρέπει να μας προβληματίσουν για τα οποία πρέπει να έχει κάθε σκάφος που αλλιεύει εις τρόπον ώστε να αποφεύγει την υπεραλίευση και να κάνει οτιδήποτε το οποίο είναι εναρμονισμένο σε αυτό το οποίο λέμε μεταρρύθμιση κοινωνικής αγροτικής πολιτικής, ε, πολιτικής το οποίο είναι ε, ένας ιονίνο πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να πάρει τον χαρακτήρα της πλήρους εξειδίκευσης, διότι αν πάμε στην πλήρη εξειδίκευση νομίζω ότι θα χάσουμε την έννοια της ε, αλληλείας σαν σύνολο σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και θα είμαι ε, διαθέσιμος κάθε παρατήρησή τους να τη συμπεριλάβω μέσα στην εκθέση μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. 15 Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Αλλασίες Υποθέσει και την Αλία. Ε, σε αυτό το θέμα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσει ο κύριος Καντέκ ε, την πρότασή του. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα θα σας προτείνω ένα χρονοδιάγραμμα. Όπως ξέρετε, έχουμε έναν κοινό κανονισμό, συζητείται ένας κοινός κανονισμός για όλα τα ταμεία και θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιοι κοινοί προσανατολισμοί. Ο κανονισμός κοινών διατάξεων προβλέπει προϋποθέσεις που θα ισχύουν για όλα τα ταμεία, όπως και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και ένα κοινό χρονοδιάγραμμα Επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλία δεσμεύεται και με τους προσανατολισμούς που έχουμε στον βασικό κανονισμό και με τον κανονισμό που έχει να κάνει με την κοινή οργάνωση της αγοράς. Γι' αυτό το λόγο προτείνω ότι στο δεύτερο εξάμεινο του έτους θα πρέπει να εγκριθεί ο κανονισμός για το, η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλία, γιατί θα πρέπει να ακολουθηθεί όλη η διαδικασία με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές και θα πρέπει παράλληλα να ασχοληθούμε και με τον κανονισμό κοινών διατάξεων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τι Θαλάσσιε Υποθέσει και την Αλία εξαρτάται επίση από το πολιετέ δημοσιονομικό σχέδιο από το 2014 και μετά, επομένω εντάσσεται στι δημοσιονομικέ προοπτικέ, μελλοντικέ δημοσιονομικέ προοπτικέ. 27 Φεβρουαρίου, λοιπόν, σα προτείνω να γίνει μια γενική ανταλλαγή απόψεων. Στι 24 Απριλίου, παρουσίαση του εγγράφου εργασία και ανταλλαγή απόψεων. Στι 30 Μαου, μία ακρόαση για το Ταμείο αυτό, οργανωμένη από την, Ευρωπαϊκή, από την Επιτροπή Αλίας, 19 Ιουλίου ανταλλαγή απόψεων, 19 Ιουλίου ανταλλαγή απόψεων, το Σεπτέμβριο παρουσίαση 9 Οκτωβρίου ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες και στις 6 Νοεμβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή Αλίας. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο σας προτείνω και αυτό έχω να σας πω μόνο αυτή τη στιγμή, γιατί όπως σας είπα ο βασικός κανονισμός δεν έχει προχωρήσει ακόμα, επομένως και εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πολύ ωραία. Κυρία Φράγκα, θέλετε να πείτε κάτι για το χρονοδιάγραμμα. Θέλει να μιλήσει κάποιο για το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, δεν έχουμε προβλέψει συζήτηση τη ουσία. Σύντομα, κυρία Φράγα. Ναι, εγώ θα ήθελα να εκφράσω μια σκέψη. Και για τον συγκεκριμένο, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι το εξή. Το συζητήσαμε και το πρωί με την κυρία Υπουργό. Η πρόταση που κάνει η Κομισιόν για το νέο ταμείο είναι μια πρόταση όπου αποσύρονται εντελώ οι ενισχύσει του για το στόλο. Εγώ είπα ότι είμαι υπέρ ε, στο να καταργηθούν ε, αυτές οι ενισχύσεις, αλλά βέβαια το, για το πόσο θα συνεχιστούν ε, είναι μια... Δεν είναι θεμοσίε, είναι υποκρασία. όμως το μοντέλο διαχείρισης είναι αυτό που έχει τις μεγαλύτερες οικονομικές λήψεις, γιατί η μελέτη διεκτυπή τη Κομισιόν μα δείχνει ότι αν δεν τροποποιηθεί το μοντέλο διαχείριση και αν δεν κινηθούμε προ ένα πιο αποτελεσματικό οικονομικό μοντέλο, τότε θα χρειαστεί να συνεχίσουμε με τι επιδοτήσει. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε πρόβλημα αν εμείς δεν τροποποιήσουμε τίποτα από την κοινή ελευθερική πολιτική και αναφέρομαι κυρίω στο μοντέλο διαχείριση, θα πρέπει να έχουμε ενισχύσει, γιατί διαφορετικά ο στόλο δεν μπορεί να επιβιώσει. Και αυτό το λέει το impact assessment τη Κομισιόν, δεν το λέω εγώ. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα ουσίας. Δηλαδή είτε και τα δύο θα θα τροποποιήσουμε τίποτα. Θέλω να πω. Εγώ που προσωπικά υποστηρίζω να αλλάξουμε το καθεστώ των ενισχύσεων, θέλω να αλλάξουμε και το μοντέλο διαχείριση. Πρέπει να υπάρχει μια διασύνθεση και αν δεν υπάρχει τροποποίηση τότε πρέπει να έχουμε ενισχύσει για να βοηθήσουμε το στόλο. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι θέμα ουσία και πρέπει να το έχουμε υπόψη όταν θα λάβουμε αποφάσει. Μάλιστα ευχαριστούμε κύριε Φράγκα, δεν θα μιλήσουμε θέμα, για θέματα ουσία σήμερα. Θα έχουμε πολλέ ευκαιρίε το κάνουμε και θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν αν θέλει να να αφαιρθεί στο θέμα του χρονοδιαγράμματος, όχι στο θέμα του ταμείου. Ναι, κοιτάξτε, για το χρονοδιάγραμμα θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικό, καθώς η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο προετοιμάστηκε ε, από την Κομισιόν ε, μήνες μετά το βασικό κανονισμό και στο μέτρο που αυτού του κανονισμού πρέπει να θετηθεί πριν το 2014, θα προτιμούσαμε πριν από τα μέσα του 2013 για να έχουμε χρόνο να αναπτυχθούν τα επιχειρησιακά προγράμματα με τα κράτη-μέλη. Θεωρούμε ότι μπορεί να αρκεί ο χρόνο αυτό, λαμβάνοντα και υπόψη, όπω ακούσατε και από τη Δανέζα Υπουργό, η Προεδρία τη Δανία σκοπεύει να σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη συζήτηση στο Συμβούλιο, έτσι ώστε από τα σκοπιά της Κομισιόν ε, το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μας επιτρέπει να ε, μπορεί να υιοθετηθεί αυτός ο κανονισμός περί τα μέσα του 2013. Αυτό χρειαζόμαστε για να έχουμε το, το τελευταίο εξάμεινο του 2013 για να προετοιμάσουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα από τα κρατημέλη και να μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανονισμό το 2014 όταν θα πρέπει να κάνουμε την αντικατάσταση του Ταμείου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάντεκ. Ωραία, δεν θέλετε το λόγο. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο, 16. Αλία μικρή κλίμακα και παραδοσιακή ελία. και μεταρρύθμιση με τη ΣΚΑΛΠ για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ο κ. Φεραίρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ εκπώνησα ένα γράφο εργασία ε, και ελπίζω ε, να σας έχει μοιραστεί. Τώρα θα αναφέρω ορισμένα από τα σημεία αυτού του εγγράφου εργασίας ε, για να υποστηρίξουμε έτσι τη συζήτηση. Η αλία μικρής κλίμακας, ε, θα την αναφέρω από εδώ και πέρα ως μικρή αλία, για να πλουστεύσω. Το πρώτο θέμα που τίθεται και είδαμε στην προηγούμενη συζήτηση είναι το θέμα του ορισμού. Το αυτό που τελικά, τι είναι δηλαδή τελικά. Ε, αλία μικρής κλίμακας. Έχουμε ποικιλόμορφες καταστάσεις ε, στα κράτη-μέλη, όμως παρά, παρά από αυτή την ποικιλομορφία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών κοινών. Χαρακτηριστικά που μπορούμε να προσδώσουμε στην αλία μικρής κλίμακας ε, και μπορεί να υπάρχει μια συνένεση σε σχέση με αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα αναφέρω ορισμένα. Έχουμε ένα είδος αλία. που ε, με άλλους ε, τομείς που χαρακτηρίζουμε βιομηχανική ελεία, σε σχέση δηλαδή με αυτούς τους τομείς, ε, η μικρή αλεια σχετίζεται πιο ισχυρά στην κοινωνική δομή και στην οικονομική δομή των ε, παράκτιων κοινοτήτων. Σχετίζεται πιο πολύ με τις παραδόσεις και τον πολιτισμό, την κουλτούρα των κοινοτήτων αυτών. Δεύτερο σημείο, Ελία Κλίμακας. Ε, η άσκηση των δραστηριοτήτων γίνεται πιο κοντά στην ακτή και οι αλείς μένουν λιγότερο καιρό, λιγότερο χρόνο στη θάλασσα. Τρίτο, ε, έχουμε μεγαλύτερη χρήση εργατικού δυναμικού ανά μονάδα άλλη πτυχή. Συνήθως η μικρή Ελία χρησιμοποιεί πιο επιλεκτικά εργαλεία που έχουν μικρότερες επιπτώσεις από των πόρων. Άλλη πτυχή, αυτή η μικρή αλία ε, συνήθως ε, μπαίνει σε πιο απλές αλυσίδες τροφοδοσίας, ε, παίρνει το σχάρι, ε, δεν τροφοδοτεί τη μεταποίηση, τη μεταπητική μηχανή, αλλά έχουμε κατανάλωση νοπών προϊόντων και άλλα χαρακτηριστικά μπορεί να υπάρξουν. Άλλη πτυχή είναι ότι μεταξύ των αλλιεών υπερισχύουν οι μικρές επιχειρήσεις ή οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν παρά την μεγάλη ποικιλομορφία που υπάρχει, αυτό το σύνολο χαρακτηριστικών μας επιτρέπουν ε, να διαφοροποιήσουμε την αλία αυτή από τη βιομηχανική αλία, την αλία μεγάλης κλίμακας. Και αυτές οι δύο μεγάλες ομάδες ε, θα πρέπει να τύχουν διαφορετικές μεταχείρισης, θα πρέπει να ε, έχουμε μοντέλα διαχείρισης που να σέβονται τις ιδιαιτερότητές τους. Δεν ε, μπορούμε να έχουμε ένα ομοιομορφό μοντέλο, πείσουμε δύο εντελώ διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να αναλύσουμε το σύνολο των προτάσεων της Κομισιόν και να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος των προτάσεων αυτών ε, στην ε, μικρή παρακτηλία. Στην Ελία Μικρή Κλίμακα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ιδιαιτερότητε τη Ελία Μικρή Κλίμακα δεν λαμβάνονται παρκώ υπόψη στι προτάσει τη Κομισιόν. Επίσης δεν δίνεται κατάλληλη απάντηση στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλία μικρής κλίμακας. Η πρόταση της Κομισιόν ε, συνεχίζει να έχει μία προσέγγιση συγκεντρωτική ε, της ΚΑΛΠ. Ε, επίσης, ο τομέας δεν συμμετέχει στην εκπόνηση στη συζήτηση για την εκπόνηση της νομοθεσίας και το κεφάλαιο της περιφερειοποίησης δεν εγγυάται ε, αυτή την ε, εγκύτητα ε, με τους μικρούς αλείς. Και επίση για το υποχρεωτικό χαρακτήρας των μεταβάσιμων ελευτικών παραχωρήσεων ίσως ε, θα είναι το πιο σοβαρό ε, για την αλία μικρή κλίμακα Η Κομισιόν υιοθετεί και πάλι εδώ ένα ορισμό που αποκλείει τη μικρή αλία από αυτό το καθεστώς. Υιοθέτησε έναν ορισμό που είναι πολύ απομακρυσμένος από την πραγματικότητα. Υπόθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση. Έχουμε δηλαδή και το θέμα των 12 μέτρων και ο ορισμός που δεν περιλαμβάνει ένα ουσιαστικό τμήμα αυτού που πρέπει να θεωρήσουμε ως αλία μικρής κλίμακας αφενός και αφετέρου ε, δεν ε, θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα και να καλύψουμε τις ανάγκες της ελίας μικρής κλίμακας με αυτό το υποχρεωτικό σύστημα. Η Κομισιόν ε, προβαίνει σε συγκέντρωση ε, της δραστηριότητας στο τομέα για να το αποφύγουμε αυτό, για να το αποφύγει μάλλον αυτό, ε, προβλέπει αποκλεισμό των σκαφών μέχρι τα 12 μέτρα, όμως αυτό δεν αρκεί. Δηλαδή προβλέπονται κάποιες ρήτρες διασφάλισης αλλά δεν αρκούν. Γιατί ο τρόπος που λειτουργεί η ενιαία αγορά ε, δεν θα εμποδίσει να υπάρχει συγκέντρωση ε, των δικαιωμάτων αυτών στις μεγάλες επιχειρήσεις και μάλιστα θα το δούμε αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν ε, να παρεμποδίσουμε το φαινόμενο αυτό. σε σχέση με την πρόταση της κοινή οργάνωσης ε, αγοράς. Δεν απαντώνται πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η, μικρή, η αλία μικρή κλίμακας, ε, η μείωση των τιμών πρώτη πώληση, ε, επίσης η άνηση κατανομή κατά τη διάρκεια της ελισίδας Και σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και απαγορεύοντας ε, την οικοδόμηση νέων λιμενιών, νέων ε, τόπων εκφόρτωσης και πάλι δεν λαμβάνει υπόψη η Κομισιόν ε, την αλία μικρής κλίμακας και ε, την ποικιλομορφία της στα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, είσοδος νέων αλλιέων ε, στη δραστηριότητα και εγγύηση ανάπτυξη του τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίζει να αναπτύσσεται η αλλία μικρής κλίμακας Επίσης ε, υπάρχει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλίας μία διάκριση ε, της ε, Αλίας εναντί της εδωτοκαλλιέργειας ε, και γιατί θέλετε να περιορίσετε την είσοδο νέων στον τομέα. Γιατί σε πολλά κράτη-μέλη βλέπουμε ότι χρειάζεται να μπουν νέοι στον τομέα στην αλία μικρής κλίμακας. Το θέμα της ενημέρωσης και της απόκτησης δεδομένων αναφέρθηκε εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαθεσιμότητα πληροφοριών ε, είναι απαραίτητη για να λειτουργεί η διαχείριση, για να υλοποιείται η διαχείριση και αυτή η διαθεσιμότητα των πληροφοριών καθίσταται ακόμη πιο απαραίτητη καθώς η πραγματικότητα μας θέτει πάρα πολύ σοβαρές προκλήσεις ως προς τη διαχείριση και Φυσικά η διαχείριση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, επειδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διαφοροποίησεις και γι' αυτό χρειαζόμαστε τις πληροφορίες. Επίσης, ε, πρέπει να μελετούμε εξαντλητικά τα χαρακτηριστικά της αλίας μικρής κλίμακας. Πρέπει να γνωρίζουμε πού, πώς, πότε αλλιεύουν ε, τα διάφορα τμήματα του κλάδου που εμείς συμπεριλαμβάνουμε σε αυτόν τον ορισμό αλλία μικρής κλίμακας. Και φυσικά έτσι καθίσταται απαραίτητη η αύξηση των κοινοτικών προσπαθειών στη χρηματοδότηση για την απόκτηση και τη διαθεσιμότητα αυτών των πληροφοριών. Δυστυχώ ε, κάτι τέτοιο δεν καλύπτεται στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Ελίας. Έτσι λοιπόν. Ε, παρά το ότι σήμερα προβλέπει η συνθήκη διαχείριση τη ελία να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πραγματικότητα αυτό που λέγεται σε σχέση με το κόστος ορισμένων πτυχών που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση όπως απόκτηση πληροφοριών συνεχίζει ε, να ε, θέτει στα κράτη-μέλη ένα σημαντικό τμήμα του κόστους για την αποκτήση και διάθεση αυτών των πληροφοριών, ενώ εδώ θα έπρεπε να δούμε μία αύξηση και της ε, συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να βελτιώσουμε δηλαδή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Θεωρώ Αυτές οι προτάσεις θα μπουν σε ένα γράφο εργασίας που θα σας μοιράσουμε και ελπίζω να υπάρχει και ευκαιρία να συζητήσουμε περαιτέρω τα θέματα αυτά. Καταρχήν ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα υποστήριξης ε, της ε, αλίας μικρής κλίμακας σε κοινοτικό επίπεδο, να περιλαμβάνεται εκεί το ε, χρηματοοικονομικό σχέδιο, η κοινή οργάνωση αγοράς, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, που θα μας βοηθήσουν να απαντήσουμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και να μπορούμε να έχουμε βιώσιμη ελεία. Πρέπει να ε, εγγυηθούμε ε, από το νέο Ταμείο Αλίας τα απαραίτητα κονδύλια για τον εξυγχρονισμό των στόλων, να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφαλείας, πρέπει να έχουμε αηφορία σε περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο και να προσθέσω κάτι εδώ, η Κομισιόν στην πρόταση μεταρρύθμισης ε, θέτει κάποιους περιβαλλοντικού στόχου. Αυτό αναφέρθηκε και όταν συζητήσαμε την γνωμοδότηση του κ. Σαλαβράκου. Η Κομισιόν θέτει συγκεκριμένους στόχους περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όμως δεν θέτει συγκεκριμένους στόχους σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και για τον ε, τομέα της μικρής ελίας ε, που βιώνει μια τραγική κατάσταση σε πολλές χώρες ε, πρέπει να τεθούν και στόχοι αυτοί. Αυτό το πρόγραμμα στήριξης στη μικρή ελία. θα πρέπει να ε, βοηθήσει τους νέους ε, να μπουν στον τομέα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε επαγγελματική κατάρτιση, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και να αξιολογούνται οι δραστηριότητες των αλλιέων και θα πρέπει να προσδώσουμε και αξία στο ρόλο που διδραματίζουν οι γυναίκες στην αλλία και συγκεκριμένα στην αλλία μικρής κλίμακας. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε διαφοροποιημένη μεταχείριση της αλίας μικρής κλίμακας, ε, ένα της μεταχείρισης που έχουμε για τη βιομηχανική αλία και ο καλύτερος τρόπος να υπερασπίσουμε την αλία μικρής κλίμακας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση θα ήταν ένας ε, κατακαιρματισμός ε, στο χώρο των δύο ειδών αλίας κάθε, σε κάθε, κάθε κράτος μέλος ε, θα πρέπει ε, να καθορίσει ε, σε ποιες προστατευόμενες περιοχές, σε ποιες περιοχές έχουν πρόσβαση οι αλίες μικρής κλίμακας. Επίσης, θα Πρέπει να δούμε και τη συνεισφορά των ε, παράκτιων κοινοτήτων ε, στο περιβαλλοντικό, στο κοινωνικό και στο οικονομικό επίπεδο. δεν ε, θα πρέπει να αποδυναμώσουμε πολλά από τα εφιστάμενα δημόσια εργαλεία που έχουμε για να υποστηρίξουμε αυτό το τομέα. Και πριν από τη δική μου παρέμβαση ακούσαμε και τι είπε και η συνάδελφος η κυρία Φράγκα. Είναι αδύνατο να μην εξετάσουμε τη βιωσιμότητα του τομέα της αλίας μικρής κλιμικάς και της Περιδοσιακής αλίας στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ε, παράλληλα ε, σκεφτόμαστε ότι θα καταργηθούν ε, οι ενισχύσεις. Μέχρι τώρα ε, έχουμε θετικέ εμπειρίε ε, για από την Ελλήνη και και η ίδια η Κομισιόν το είπε και εμεί θεωρούμε ότι ε, πρέπει να ε, καθιερώσουμε την αρχή που έχουμε εκεί και θα πρέπει να εξετάσουμε και τη δυνατότητα διεύρυνσης ε, αυτών των 12 μιλιών που έχουμε, της αρχής των 12 μιλιών ε, και να φτάσουμε και μέχρι τις υφαλοκρηπίδες. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε τη δυνατότητα να διευρύνουμε κυρίως τις ε, άκρως απομακρυμένες περιοχές. Ίσως θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι και τα 200 μίλια όπως έχουν ζητήσει πολλές από αυτές τις περιοχές. Και προτείνουμε εδώ τη δυνατότητα να εξετάσουμε τη δημιουργία μηχανισμών έκτατου ανάγκης καθώς ε, υπάρχουν διαρθρωτικές ε, αδυναμίες στον τομέα. Ο τομέας της μικρής ελίας είναι πιο εκτεθειμένος σε εξωτερικά σοκ ή σε ε, ευνίδιες αλλαγές. Αυτή η κατάσταση σήμερα επιβαρύνεται λόγω της αστάθειας των αγορών, των χαμηλών τιμών πρώτης πώλησης και επειδή αυξάνεται το κόστος παραγωγής και το κόστος των καυσίμων. Έτσι λοιπόν προτείνουμε να εξεταστεί δυνατότητα να δημιουργήσουμε συγκεκριμένους μηχανισμούς στήριξης που θα δραστηριοποιούνται, θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση ε, συγκεκριμένων ε, περιπτώσεων όπως είναι άνοδος των τιμών των καυσίμων, ε, φυσικές καταστροφές κτλ. Επίσης η στήριξη στις, ε, ε, βιολογικές απαγορεύσεις θα πρέπει να υπάρχει και θα πρέπει να έχουμε ε, την ε, σύσταση κάποιων περιόδων ε, απαγορεύσεις της αλίας Όμως ε, θα πρέπει κατά τη διάρκεια αυτής ε, της περίοδου όπου υπάρχει απαγόρευση, βιολογική απαγόρευση, να υποστηρίζουμε τους ε, μικρούς αλείς. Σήμερα η αλία μικρής κλίμακας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και πρέπει να προσδώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο πώς θα συμμετέχουν οι μικροί αλείς στη διαχείριση και στην εφαρμογή των πολιτικών. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις επαγγελματικές οργανώσεις, τις ομάδες ε, των παραγωγών που είναι έτοιμοι ε, να επιμεριστούν την ευθύνη για την εφαρμογή της κάλψης. Σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλοι η περιορισμοί ε, της συμμετοχής των μικρών αλλιέων στα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια. Αυτό το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί και θα πρέπει να κατατεθούν κάποια μέτρα για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστούμε για τις εξαιρετικές ε, εξηγήσει. Πέντε συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Δύο λεπτά το πολύ σας παρακαλώ. Κυρία Λοβέν. Και μετά κυρία ε, Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Χωάο για την ε, παρουσίασή σου. Είμαι περίεργη όσον αφορά την πρότασή σου και την ανάλυση. Μας έδωσες κάποια στοιχεία, αλλά έχει αναλάβει μια πολύ σημαντική πρόκληση. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το θέμα, όπως είπαμε όλοι. Ε, το να ορίσουμε δηλαδή ποια αλληλεία είναι πράγματι μικρής κλίμακας. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι δεν είναι πάντα τόσο προφανές. Για μένα πιο σημαντικό είναι ε, η αλληλεία να είναι βιώσιμη και μερικές φορές ε, δυστυχώς ε, η υποβάθμιση του ε, θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε υπερβολική ικανότητα της, ακόμα και της αλίας μικρής κλίμακας. Έτσι λοιπόν μπορεί και η αλία μικρής κλίμακας να είναι βλαβερή για το θαλάσσιο περιβάλλον και σίγουρα θα πρέπει να μειωθεί σε, σε πολλές περιοχές. Αποτελεί λοιπόν και αυτό πρόκληση. Πώς θα το πετύχουμε αυτό. Ένα στοιχείο που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι αυτό που είπες για την συνδιαχείριση. Οι αλλοίς μικρής κλίμακας ε, να έχουν και αυτοί μια φωνή που συχνά δεν ε, ε, νιώθουν ότι εκπροσωπούνται από τις οργανώσεις παραγωγών. Υπάρχουν δυνατότητες στον λεγόμενο άξονα 4 όπου ε, έχουμε εκατοντάδες προγράμματα σε όλη την Ευρώπη που κατά μέσον όρο έχουν λάβει 3 εκατομμύρια ευρώ ανά πρόγραμμα. Μπορούν έτσι να προσθέσουν αξία στα αλλιεύματά τους, μπορούν να εκπαιδευτούν, μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους τομείς πέρα από την αλληλεία. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα, και θα ήθελα να το τονίσω αυτό, ε, υπάρχει και η δυνατότητα ε, τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν από αλληλείς μικρής κλίμακας. Εάν ενωθούν μπορούν να δουν πώς μπορούν να ε, οργανώσουν την συνδιαχείριση και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους σε εποχές πιθανότατα ιδιωτικοποίησης της θάλασσας. Θα, ε, ε, ελπίζω αυτό να τονιστεί επίση στην εκθεσή σου όσον αφορά την ε, προστιθέμενη αξία των αλλιευμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους αλλιεί μικρής κλίμακα. Δεν μπορούν να επιβιώσουν αποκλειστικά με την αξία των αλλιευμάτων τους. Η προστιθέμενη αξία αποκτάται από όλους τους μεσάζοντες θα πρέπει οι ίδιοι να βγάζουν περισσότερα χρήματα από την αλληλεία και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Επίσης, ε, όσον αφορά την αρχή της ευέλτιστης διαθέσιμης πρακτικής ε, για όλη την αλληλεία, θα πρέπει να εφαρμοστεί και για τους αλληλείς μικρής κλίμακας. Εάν, ε, έχουν, εάν είναι καλύτεροι στον άλλη, έχουν κάποιο συγκεκριμένο απόθεμα, να έχουν πρόσβαση προτεραιότητας. Ευχαριστώ κύριο Κάλαχερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προέρχομαι από την επαρχία της Ιρλανδίας με πολλά νησιά στην εκλογική μου περιφέρεια. Δεν θα υποβάθμιζα ποτέ λοιπόν την αξία της αλίας μικρής κλίμακας και ε, ο Ζωάς στην αρχή της ε, παρουσίασή του αναφέρθηκε στην κοινωνική σημασία, την ε, οικονομική, την ε, παράδοση. Ε, λόγω του περιορισμένου μεγέθους των σκαφών δεν μπορούν να απομακρυνθούν πολύ από την θάλασσα. Μπορεί να είναι δηλαδή επικίνδυνο το να αλλιεύουν εκτός των κλειστών περιεχών. Ε, χρειάζονται πολύ ε, εργασία τα μικρά σκάφη, έχουν δύο ή τρία άτομα και τι κάνουν, βοηθάνε στην ε, επιβίωση οικογενειών σε πιθανότατα τις πιο φτωχές υπαίθριες περιοχές της Ευρώπης. Παρέχουν απασχόληση σε περιοχές όπου δεν υπάρχει εναλλακτική πηγή απασχόλησης. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τα απαραίτητα χρήματα για γεωργικά προγράμματα, για παράδειγμα. Φυσικά μπορούν να απασχοληθούν σε μεγαλύτερα σκάφη και ε, ενδεχομένως με επενδύσεις να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, δεν εργάζονται 52 εβδομάδες ε, την, ε, το χρόνο, 7 ημέρες τη εβδομάδα; Θα μπορούσε εκτός εποχής να απασχοληθούν αλλού. Πιο σημαντικό είναι ότι έχουν ε, ελάχιστο ή ε, καθόλου αντίκτυπο ε, στα αποθέματα. Αν κάποιος υπονοεί ότι είναι υπεύθυνοι για την εξάντληση των αποθεμάτων, αυτό δεν είναι αλήθεια. Ούτε θα πρέπει να τους κρίνουμε με τον ίδιο πύχη με τα μεγάλα σκάφη. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα νωρίτερα για το κείμενο της ανακοίνωσης. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι υπήρχε παραδοσιακά. Τα σκάφη 15 μέτρων και οι άνθρωποι που αλλιεύουν στα μικρά αυτά σκάφη είναι θαραλέοι, διότι ουσιαστικά διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Κλείνοντας, να πω ότι δεν θα πρέπει να ε, υποτιμήσουμε την αξία τους και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διατηρήσουμε την αλήθεια αυτή. Ε, κινδυνεύω να επαναλαμβάνομαι, με κίνδυνο να επαναλαμβάνομαι να πω ότι δεν είναι εκείνη υπεύθυνη για την εξάντληση των αποθεμάτων. Ε, θα προσλέπουμε στην περαιτέρω συζήτηση όταν θα είναι διαθέσιμο το έγγραφο εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρόντουστ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν ε, μίλησα πολύ σήμερα επειδή η φωνή μου δεν ε, τα πάει πολύ καλά και ούτε εδώ ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Φερέιρα. Στην κοινή αλλιευτική πολιτική η, η αλληλεία μικρής κλίμακας δεν λαμβάνει τη θέση που της αξίζει. Πιστεύω ότι ε, το έργο του κυρίου Φερέιρα καθώς και η έκθεση που θα υποβάλει τελικά θα είναι σημαντικό έγγραφο εργασίας ε, για μας. Ε, γι' αυτό τον ευχαριστώ θερμά. Θα πρέπει καταρχήν να βρούμε έναν ορισμό. Ο δικός μου ορισμός δεν έχει να κάνει με το μήκος των σκαφών. Συνδέεται περισσότερο επικεντρώνεται περισσότερο στον όγκο των αλλιευμάτων. Για μένα είναι σημαντικό να καταστήσω σαφές το εξή. Η αλληλεία μικρής κλίμακας ε, δεν είναι πάντα καλή. Μπορεί να υπάρχουν οικολογικά προβλήματα αλλά και οικονομικά και γι' αυτό θέλουμε να φροντίσουμε όχι μόνο να έχουν ευκαιρίες για επιβίωση αυτές ε, αυτά τα σκάφη μικρής ε, κλίμακας, αλλά να έχουν και δυνατότητες ε, εκπαίδευσης ε, και κατάρτισης. Ε, και τελευταία πρόταση, χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε αποφασίσει να συζητήσουμε μαζί τα τρία βασικά τιμία, το γεωργικό, τα και το περιφερειακό, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν μέτρα μετεκπαίδευση. Ευχαριστώ. Grazie Presidente, io sono un nuovo componente di questa ε, Εγώ αποτελώ νέο μέλο ε, τη Επιτροπή και προέρχομαι από την ε, Νότια Ιταλία και έχουμε 740 χιλιόμετρα ακτής πάνω από 740 χιλιόμετρα ακτής ε, και θέλω να χαιρετήσω ε, τα όσα είπε ο κύριος Φερέιρα γιατί με απασχολούν και μένα πολύ προσωπικά. Βέβαια ε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη ε, διάθεσή μας τώρα και μόλις λάβαμε και το κείμενο εργασίας και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο μέλλον και να κάνουμε περαιτέρω σχόλια. Αλλά θα ήθελα να φερθώ σε κάποια σημεία. Η Ηλία της μικρή κλιμακα ε, έχει πραγματικά πολύ στενή σχέση με την ε, επικράτεια. Με, ε, και αυτό θα πρέπει να το προωθήσουμε να του προσδώσουμε αξία, γιατί πολλές φορές έχουμε οικογενειακές επιχειρήσεις, έτσι λοιπόν πρέπει να προσδώσουμε αξία και στις επιχειρήσεις αυτές. Κάτι που με απασχολεί εμένα περισσότερο, που μου είναι πιο οικείο, είναι αυτό που ανέφερε ο κύριος Φερέιρα και έχει να κάνει με την είσοδο των νέων στον τομέα. Δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσουμε και να ευνοήσουμε τους νέους ελλείς και θα πρέπει να τους προσδώσουμε καλύτερη κατάρτιση, ε, επαγγελματική κατάρτιση και εγώ, να σας πω, για πολύ καιρό ήμουν ε, ε, σύμβουλος ε, στη δική μου περιφέρεια, στον τομέα της γεωργίας και ασχολήθηκα με το θέμα της κατάρτισης και είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Και θα πρέπει να προσανατολίσουμε περισσότερο το τομέα προς την αγορά για να καταργήσουμε τις ενισχύσεις. Και Θέλω να ρωτήσω μήπως ε, θα μπορούσαμε να έχουμε και κατά νου την ε, ιδέα ε, της αλίας ως τουριστική δραστηριότητα. Υπάρχουν κάποια τέτοια σκάφη. Συγγνώμη, η πρώτη φορά, Πρόεδρε, παίρνω το λόγο. Άλλοι μίλησαν περισσότερο από μένα, οπότε δώστε μου λίγο χρόνο. Να δούμε λοιπόν και το θέμα αυτών ε, των ε, σκαφών. Και κάτι άλλο που δεν πρέπει να υποτιμούμε είναι οι φυσικές καταστροφές. γιατί δίνονται, πρέπει να δίνονται επαρκείς ενισχύσεις έτσι ώστε οι αλείς που αντιμετωπίζουν ε, πολλές δυσκολίες σήμερα θα πρέπει να τους βοηθήσουμε γιατί διαφορετικά ο τομέας θα πάψει να θα πεθάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Φερέιρα για το εργαστήριο. Απλώ ήθελα να σα πω ότι εγώ στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτική θα είμαι ε, η συγγήτρια για το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν ε, θα αναφέρουμε ότι ε, θέλουμε να συμπεριληφθούν θαλάσσιοι οργανισμοί. Η αλία θαλάσσιων οργανισμών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ 100% με αυτά που είπε ο κύριος Φερέιρα. Νομίζω ότι ο κοινός μας στόχος είναι να καταστήσουμε την μικρή αλία πιο αποτελεσματική, πιο λειτουργική. Θα πρέπει σε αυτή να βασιστεί η μελλοντική κοινή αλληλευτική πολιτική. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον ανταγωνισμό που έρχεται από τις μεγάλες εταιρείες. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες προκειμένου η μικρή αλληλεία να είναι λειτουργική, να μπορεί να ανταγωνιστεί οι μεγάλες εταιρείες, να μπορεί να επιζήσει. Όσον αφορά επίσης τη βιώσιμη αλεία, πιστεύω ότι η αλία μικρής κλίμακος ουσιαστικά συμβάλλει πολύ περισσότερο στη βιωσιμότητα της αλίας, γιατί οι παραδόσεις βασικά των παλαιών αλίεων περνάνε στις νέες γενές και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται σεβαστή μία κάποια συνέχεια επαγγελματική αν θέλετε. Οι μικρές αυτές αλιευτικές εταιρείες εκτιμούν ιδιαίτερα την αλία, νοιάζονται για τη βιώσιμότητά της, ακριβώς επειδή ζούνε από αυτήν. Στις μεγάλες εταιρείες δεν υπάρχει η συναισθηματική αυτή σχέση. Ευχαριστώ κυρία Πατράου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμείς ε, εδώ στην Επιτροπή Αλίας ε, πάντοτε ομόφωνα είμαστε υπέρ ε, της αλίας μικρής κλίμακας και όσο προχωρά ο διάλογος ε, ε, αναδύονται και διάφορες ε, ιδέες. Θέλω να αναφερθώ εγώ σε τρία σημεία. Αρχίσαμε να ακούμε, να, να ε, πολλές φορές ότι η μικρή αλία ε, ουσιαστικά ε, α, μειώνει την, τα αποθέματα. Όμως πρέπει να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι λόγω των εργαλείων που χρησιμοποιούν οι μικροί Ελλεί δεν υπάρχει μεγάλος αντίκτυπος στα αποθέματα. Έτσι λοιπόν γι' αυτό πρέπει να έχουμε και έναν κατάλληλο ορισμό της ε, αλίας μικρή κλίμακα. Επίσης, θέλω να φερθώ στην απουσία ενισχύσεων για τους μικρούς Αυτό μα ανησυχεί, γιατί ε, η αλία μικρή κλίμακα είναι πολλά περισσότερα από την ε, αλίευση ψαριών και τη θέση του σε εμπορία. Μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία ε, έχει να κάνει με τη ζωή στις παράκτιες περιοχές και πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Και τρίτη πτυχή, είμαι κατά τις πρώτες της Κομισιόν για τις ε, ατομικές μεταβάσιμες ελευτικές παραχωρήσεις, ε, να καταστεί δηλαδή αυτό το καθεστώς υποχρεωτικό και θέλω να ρωτήσω, σε περιοχές, σε ζώνες όπως παραδείγματος χάρη οι άκρως απομακρυσμένες περιοχές, πώς ε, τα σκάφη της ε, αεραστεχνικής αλίας ε, θα τα ε, αντιμετωπίσουν, πώς θα τα μεταχειριστούν αν έχουμε ένα υποχρεωτικό σύστημα των μεταβιβάσεων παραχωρήσεων. Έχουμε λοιπόν αυτού του κινδύνου που θα μπορούσαν να αναπλήξουν αυτή τη δραστηριότητα της μικρής Ελία. Ευχαριστώ, επόμενο ομιλητή. Ναι, πολύ γρήγορα. Δύο σκέψει. Και προτάσεις εργασία ε, στον κύριο Φερέιρα, που έχει κάνει μια εξαιρετική έκθεση. Καταρχήν, εγώ θα προσπαθούσα να, να αξιολογήσω και το θέμα της τοπικής αγοράς. Ο κύριος ανταγωνιστής ε, είναι η ψυχαγωγική αλληλεία για ψυχολογικούς λόγους. Και νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε και θα ήταν χρήσιμο ε, να βάλετε και αυτό το στοιχείο στην έκθεσή σας, έτσι ώστε να κατανοήσουμε ε, καλύτερα ποια θέση πρέπει να λάβουμε. Δεύτερο θέμα που αφορά και το βασικό κανονισμό, αλλά αφορά συνολικά και τη νέα πολιτική που προσπαθούμε να συστήσουμε. Κυρίως για την αλία μικρής κλίμακας ε, γίνεται στρατική της θάλασσας ως πόρο. Ε, ως ε, Προσπαθώ να εξηγήσω. Εμείς έχουμε μία παθητική ε, αντιμετώπιση, μία παθητική στάση ό,τι αφορά τη διαχείριση των θαλάσσιων χώρων. Πολλές φορές η αλία μικρής κλίμακας ε, ουσιαστικά ε, χρησιμοποιεί αυτές τις περιόδους απαγόρευσης ε, για να αμείβονται οι αλείς, αλλά και να μπορεί και η θάλασσα να ανανεώνει τους πόρους της και να μπορεί να, να παράγει βιομάζα. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για τη μικρή αυτή αλία να αναπτύξουμε αυτή αυτή τη λογική και να καθορίσουμε κάποιους χώρους που δεν είναι μόνιμες προστατευόμενες περιοχές, αλλά χώρους οι οποίοι για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους ε, και για μήνες ε, ή για χρόνια μπορεί να επιβάλλεται εκεί ε, μία no-fish area, δηλαδή όπου δεν θα υπάρχει αλία, λευτική δραστηριότητα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Γιατί αν δεν ξεκινήσουμε από μια απαραίτητη προπόθεση και αυτό αφορά και την παράκτια αλία και την αλία μικρής κλίμακας. Αν εμείς δηλαδή δεν επιτρέψουμε στη θάλασσα ε, να αναπτύξει την ικανότητα παραγωγής της, πιθανότητα θα πρέπει μόνο ε, να διαχειριζόμαστε τις εξόδους από αυτό το τομέα. Όμως, εγώ πιστεύω ότι μια δραστηριότητα που ε, περιλαμβάνει τέτοιε δραστηριότητε, που θα περιλαμβάνει τέτοιε δραστηριότητε, μπορεί να μα βοηθήσει στην ανάπτυξη τη Αλία. Μάλιστα, να δώσουμε το λόγο στον πρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομο. Πιέζει και ο χρόνο. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρωτοβουλία σα αυτή και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος συναδέλφου μου που έπρεπε να πάει σε μία άλλη συνεδρίαση. Όπως είπαμε όμως και σήμερα το πρωί, η αλία μικρής κλίμακος είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς για την αλία αυτή. Δεν θα επισέλθω αυτή τη στιγμή σε λεπτομέρειες, δεν θα μιλήσω για τον ορισμό ή για επιμέρους στοιχεία του καθεστώτος. Καταγράφουμε πάντως όλες τις ιδέες, όλες τις προτάσεις που κάνετε και προσβλέπουμε στην έκθεση η οποία θα υποβληθεί από την Επιτροπή σας. Να φερθώ σε ένα-δύο σημεία τα οποία ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πιστεύω ότι πρέπει να διευκρινιστούν. Πρώτον, όπως σας είπα, εισάγουμε ένα νέο καθεστώς για την αλία μικρής κλίμακος. Το έχουμε ήδη κάνει αυτό στα πλαίσια του νέου καθεστώτος επιτήρησης, παρακολούθησης. Ε, λαμβάνουμε υπόψη όλες τις δαπάνες που υφίσταται το τομέας αυτός για την συμμόρφωση και έχουμε και κάποιες ριζοσπαστικές αλλαγές όσον αφορά τη διαχείριση των στόλων. Στη διαχείριση αυτή των στόλων αποκλείουμε τα μικρά σκάφη, τον στόλο της μικρής αλίας, δεν συμμετέχουν δηλαδή στα προγράμματα μείωσης του στόλου και θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ σημαντική προσαρμογή η οποία γίνεται υπέρ της αλίας μικρής κλίμακας. Θα μπορούσα να αφαιρθώ και σε άλλα ζητήματα. Τα περισσότερα πάντως που ακούστηκαν σήμερα βρίσκουν μια κάποια θέση στην πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλία. Θεωρούμε ότι μπορεί να βελτιωθεί πολύ η εκπροσώπηση των ε, στόλων μικρής ε, αλίας και προβλέπουμε επίσης ότι θα υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις αλίας και έχουμε και συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξη στα πλαίσια της αγοράς για την, αληφτία, για την αλία αυτού του είδους. Όλα αυτά τα ζητήματα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης που θα κάνουμε. Προσβλέπουμε λοιπόν στη μελλοντική συζήτηση που θα έχουμε για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για την αλία μικρής κλίμακος. Ευχαριστούμε κύριο Φερέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους και τα σχόλιά τους. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο για να αφερθώ σε κάθε ένα από τα θέματα που τέθηκαν εδώ, αλλά μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι τα σημείωσα όλα. Θέλω βέβαια να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα που αναφέραν οι συνάδελφοι, που έθιξαν οι συνάδελφοι. Το θέμα του αντικτύπου της αλληλίας μικρής κλίμακας ε, υπόθηκε όταν κάτω συνεισφέρει για να προσδιορίσουμε την έννοια της αλληλεία μικρή κλίμακα είναι ότι ε, ο αντίκτυπο του σπόρου είναι σχετικά μικρός συγκριτικά ε, με άλλου ε, τομεί του κλάδου. Έτσι λοιπόν, ακριβώς για αυτό το θέμα, ε, το ότι αν υπάρχει αντίκτυπος, δηλαδή σοβαρός ε, της μικρής αλίας στους σπόρους, δεν θα πρέπει να το παραβλέψουμε αυτό και γι' αυτό αναφέρθηκα στο ότι πρέπει να έχουμε διαθέσιμες πληροφορίες για το πού, πώς, πότε. Αυτές οι γνώσεις ε, είναι σημαντικέ. Αυτή η ακτινογραφή είναι πολύ σημαντική γιατί εμεί δεν μπορούμε να μιλάμε για πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Αυτό ήταν το πρόβλημα που είχαμε μέχρι σήμερα επειδή ασκούμε ε, συγκεντρωτική διαχείριση από τι Βρυξέλλε. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώ συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν, αυτό το θέμα της βελτίωσης των πληροφοριών είναι ουσιαστικό ζήτημα. Και φυσικά εμείς ε, πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες ε, και αυτό ε, θα πρέπει ουσιαστικά να έχει και να συνδέεται και με το θέμα των χρηματοοικονομικών πόρων. Τώρα το θέμα της υπερβολικής ικανότητας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Συχνά η Κομισιόν μας παρουσιάζει πολύ γενικούς ορισμούς ε, για την υπερελίευση, για την υπερβολική ικανότητα. Εμείς όμως πρέπει να ξέρουμε ακριβώς που υπάρχει υπερβολική ικανότητα, για ποια είδη αλίας, για ποια σκάφη. Δυστυχώς ε, δεν εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Όμως θα πρέπει ε, φυσικά η ελευτική ικανότητα να ε, προσαρμοστεί και στους υφιστάμενους σπόρους. Το πρόβλημα αυτό μπορούμε να το προσεγγίσουμε με δύο τρόπους. Δεν ε, πρέπει να βλέπουμε μόνο την ποσότητα, αλλά και την ποιότητα του στόλου. Τι κάνει η Κομισιόν, βλέπει απλά την, την, ποσότητα. Και ουσιαστικά μέσω του συστήματος των μεταβέσιμων λευτικών ε, παραχωρήσεων ε, έχουμε μία συγχώνευση και τελικά ε, θα περιοριστεί η ελευτική ικανότητα. Όμως ε, τελικά τι θα γίνει. Ε, μπορεί παραδείγματο χάρη να καταργήσουμε ε, είδη αλίας ε, που θα είναι τα λιγότερα ανταγωνιστικά όμως εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε και άλλες πτυχές ε, μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε τους τομείς του κλάδου που είναι ε, πιο αηφόροι περιβαλλοντικά και οικονομικά. Δηλαδή πρέπει να δούμε και την ποιότητα, γιατί εδώ τελικά διατηρούμε τις επιχειρήσεις που είναι πιο αηφόρες από οικονομική σκοπιά, αλλά δεν είναι απαραίτητα αηφόρες από κοινωνική περιβαλλοντική σκοπιά. Και αυτό το βλέπουμε ότι έγινε σε χώρες όπου εφαρμόστηκε το σύστημα των μεταβάσιμων λευτικών παραχωρήσεων το θέμα που ανέφερε η κυρία Λόβιν για τη βελτίωση των αποδόσεων, ε, για την ε, βελτίωση των εσόδων, ε, να έχουμε δηλαδή πιο δίκαιη κατανομή. Αναφέρθηκα και εγώ σε αυτό. Επίσης και ο κύριος Σπυρίλο αναφέρθηκε στο θέμα της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων. Το προσεγγίζει αυτό και η Κομισιόν. Ε, στο Ταμείο ελία, στην πρόταση του Ταμείου Ελία. Αυτή τη δραστηριότητα θα πρέπει να τη δούμε ω τμήμα τη ελευτικής δραστηριότητα και όχι ω υποκατάστατο τη ελευτικής δραστηριότητα, Έτσι δηλαδή όπως το έχει σκεφτεί η Κομισιόν, όλες, σε όλες τις δραστηριότητες ε, ε, μπορούμε ε, να έχουμε συμπληρωματικές δραστηριότητες. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ότι θα δοθεί τέλος στην αλία μικρής κλίμακας που, έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή στις παράκτητες περιοχές. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα, αλλά δύο ακόμη σχόλια θα κάνω για τον κύριο Μιλάν, για τις ε, τοπικές αγορές και για την ψυχολογική αλία και για το ότι μπορεί ίσως να πρέπει να αξιολογήσουμε και τον αντίκτυπο αυτού του είδους της ψυχολογικής ελείας και, τι, ε, και πώς μπορεί να ανταγωνίζεται την αιλία μικρής κλίμακας. Και φυσικά δίνουμε πάντα πολύ μεγάλη σημασία στο να δούμε ε, πώς, ε, ποιος συναγωνισμός υπάρχει μεταξύ ελίας και άλλων δραστηριοτήτων, πώς χρησιμοποιείται η θάλασσα με πολλαπλούς τρόπους. Ε, αυτά δεν υπήρχαν στην πρώτη εκθεσή μου, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον θα τα συμπεριλάβω στην έκθεση. Και επίσης για τον πιθανό ορισμό των προστατευόμενων περιοχών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα διαχείρισης, ε, ότι πρέπει να γίνεται διαχείριση εκ του σύνεγγυς όπως εμείς ε, ζητάμε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να, είναι, να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους και φυσικά και ο ίδιος ο τομέας πρέπει να συμμετάσχει στον καθορισμό των μέτρων αυτών. Και για να επανέλθω στο θέμα τουρισμού, Τη ολίας μικρή κλίμακα. Ε, αναφέρθηκαν διάφορα κριτήρια, εγώ αναφέρα τα διάφορα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και έχουμε ένα σύνολο τέσσερα κριτήρια που δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν ε, θα πρέπει να τα περιβλέψουμε. Πέρα από το θέμα του αντικτύπου των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο θαλάσσιο οικοσύστημα, Έχουμε και το θέμα των χαρακτηριστικών ε, της οικονομικής ε, μονάδας και της σύνθεσης ε, του πληρώματος. Επίσης υπάρχει και το θέμα του τελικού προορισμού των ηχθείων. Αναφέρθηκαν και θέματα που έχουν να κάνουν φυσικά και με το μέγεθος του σκαφών. Νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη. Και επίσης είναι σημαντικό και αυτή η προοπτική υπάρχει και στην Πράσινη Βίβλο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό ορισμό να είναι αρκετά ευέλικτο για να λάβει υπόψη τη μεγάλη ποικιλομορφία που υπάρχει στα διάφορα κράτη-μέλη. Μάλιστα, να περάσουμε στο σημείο 17. μας μένουν μόνο 25 λεπτά για τέσσερα θέματα. Έτσι λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και ως γενικό κριτήριο να πω το εξή. Από εδώ και πέρα έτσι θα λειτουργούμε. Στην αρχή κάθε σημείου Όποιο θα χρησιμοποιήσει το λόγο να θέλει να να το ζητήσει, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε το χρόνο. Αν δίνω περισσότερο χρόνο, γιατί μόνο δύο μου έχουν ζητήσει αρχικά το λόγο και μετά παίρνουν το λόγο 6-7, εξαντλεί το χρόνο. Έτσι λοιπόν από την αρχή όποιο ε, θέλει το λόγο να το δηλώνει για να μπορούμε να περιορίζουμε και το χρόνο. Κύριε Μιλάνα, έχετε το λόγο. για την απαλλαγή του 2010 γενικώ προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Πρόκειται για μία γνωμοδότηση ε, όπως ε, ξέρετε, μπορέσαμε να αξιολογήσουμε θετικά την παρέμβαση της Επιτροπής ε, αλλά και της παρουσίας του Ελεκτικού Συνεδρίου κατά τη σύνταξη των γράφων εργασία δεν έχουν αλλάξει πολλά από τότε. Απλώς θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία ζητήματα που υπάρχουν σε αυτή την σελίδα, σε αυτή τη γνωμοδότηση. Καταρχήν ότι το συνολικό ποσοστό εκτέλεση του προϋπηγισμού είναι 27,20% και είναι θετικό, ε, το, θετικά τα στοιχεία αυτά σε σχέση με το σύνολο των εξόδων της Ένωσης. Υπήρξε ε, ε, ουσιαστικά μια πολύ χαμηλή εκτέλεση για το κεφάλαιο 11.2 που αφορά τις ελευτικές αγορές και κυρίως ό,τι αφορά την εκτέλεση των προγραμμάτων ελίσεων για τις ε, ιδιαίτερα αποκεντρωμένες περιφέρειες, ε, η Κομισιόν ε, μας διαβεβαίωσε ότι έγινε ανάκτηση αρχές του επόμενου έτους. Το δεύτερο μικρό θέμα που πρέπει να προσέξουμε αφορά ουσιαστικά ε, μία έρευνα που λαμβάνει η χώρα σε σχέση με μία ε, επένδυση στην Γερμανία. Δηλαδή υπάρχει καθυστέρηση τέλος του προγράμματος ε, από το 2001. Και φαίνεται ότι τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο. Η Κομισιόν μας έδωσε κάποια στοιχεία που θα επιτρέψουν τελικά στην Κομισιόν να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, αυτό τον έλεγχο. Και τελευταίο θέμα, έχουμε εισαγάγει ένα μικρό σχόλιο στο σημείο 7. Εγώ ήθελα να διαφοροποιήσω σε σχέση με τις δαπάνες για τις ελευτικές συμφωνίες, ε, θα ήθελα να διαφοροποιήσω τη φωνή που αφορά ε, ε, τη διαστηρά εμπορική διάσταση από την ε, διάσταση που έχει να κάνει με την τομεακή στήριξη, δηλαδή το 72% των δαπανών έχουν να κάνουν με την εμπορική διάσταση, ενώ το 28% έχει να κάνει με τη στήριξη του τομέα. Και ως τελευταίο αίτημα, Έχουμε θέσει στη γνωμοδότηση την απέτηση το ελεκτικό συνέδριο στο στάδιο αυτό της μεταρρύθμισης της ΣΚΑΛΠ ε, να ε, παρουσιάσει κάποια έκθεση σε σχέση με την ποιότητα των δαπανών και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μας βοηθήσει όταν θα συζητήσουμε επί της και ξέρετε έχουμε ε, τη διαστηρίξει και με τη στήριξη αυτή γίνεται πολιτική. Έτσι λοιπόν είναι σημαντική και αυτή η συνεισφορά του ελεκτικού συνεδρίου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τζέρεμι από την Γραμματεία που στάθηκε στο πλευρό μου γιατί χωρί αυτόν σίγουρα δεν θα μπορούσαμε ούτε να διερευνήσουμε τόσο ει βάθο ε, την ανακοίνωση και πόσο μάλλον να κάνουμε αυτές τις προτάσεις ε, που βλέπετε στο έγγραφο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Μιλάνα. Δεν ζητά κανείς το λόγο, Επομένω από την Κομισιόν έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για την γνωμοδότηση αυτή. Να αναφερθώ σε δύο σημεία. Πρώτον, οι επενδύσει στη Γερμανία. Να ενημερώσω την Επιτροπή σας ότι ακόμα και τη στιγμή αυτή που μιλάμε, η Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων δίνει την έγκριση προς τις γερμανικές αρχές και θα καταφέρουμε να καταλήξουμε κατά αυτόν τον τρόπο σε ένα αποτέλεσμα όσον αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου. Αναφερθώ έπειτα στην παράγραφο 8 της γνωμοδότησης, όπου εδώ πέρα γίνεται μία πρόταση ότι οι πληρωμές της τομεακής στήριξης θα πρέπει να κάνει με την πρόσβαση στους πόρους αρκεί να έχουν επιτευχθεί κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την τομεακή στήριξη. Προσπαθήσαμε να, διατη... να ξεχωρίσουμε, να διακρίνουμε την τομεακή στήριξη σε σχέση με την πρόσβαση. Επομένως, άλλη είναι η πληρωμή για την πρόσβαση και άλλη πληρωμή για την τομεακή στήριξη και το κάνουμε αυτό έτσι ώστε σε περίπτωση που δεν έχουμε καλές επιδόσεις στις τομεακές στηρίξεις, τότε αυτό να μην χρειαστεί να καταβληθεί ως ποσό στα πλαίσια μιας, ενός κοινού μηχανισμού πληρωμών. Θεωρούμε όμως ότι αν ακολουθηθεί η πρόταση που γίνεται στο σημείο 8, πολλές χώρες θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή, τα σκάφη του κράτους μέλου θα αλλιεύουν, αλλά αν δεν έχουν καλές επιδόσεις μετά την τομεακή στήριξη, ουσιαστικά θα μειωθεί και η υποστήριξή τους. Δεν θα θέλαμε να δούμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα, κύριε Μιλάνα, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, Όχι. Εγώ επιβεβαιώνω αυτό που υπόθηκαν και είμαι ικανοποιημένο ε, που ε, αποσαφηνίζεται και το θέμα με τη Γερμανία. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνω όσα αναφέρονται στο σημείο 8 έτσι όπως το έχουμε προσδιορίσει γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό. Και κοιτάξτε μπορεί να τροποποιηθεί ε, αυτή η γνωμοδότηση μέχρι τις 27 Ιανουαρίου έχετε και προθεσμία να στείλετε και τροπολογίες. Μάλιστα 27 Ιανουαρίου λοιπόν το μεσημέρι προθεσμία και θα έλεγα τώρα να πάμε στο σημείο 18 γιατί από ό,τι βλέπω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σεβαστούμε το χρόνο και έτσι λοιπόν προτείνω το σημείο 20 της ημερησίας διάταξης ε, να λάβει τη θέση του 26 που έχουμε αφαιρέσει. Έτσι λοιπόν αντί για το σημείο 26 τότε θα συζητήσουμε το 20 αν συμφωνείτε. Γιατί διαφορετικά έχουμε 15 λεπτά για να δούμε τρία θέματα και θα είναι αδύνατο και θα ήθελα να έχουμε κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας γιατί είναι αρκετά σημαντικά αυτά τα θέματα. Συμφωνείτε? Λοιπόν, το σημείο 20 λοιπόν θα γίνει σημείο 26 στην ημερησία διάταξη και θα το δούμε αύριο. Συνεχίσουμε με τα 18, απελαγή του 2010, κοινωνική υπηρεσία έλεγχου της Ελίας. Ο κύριος Χατζημαρκάκης έχει το λόγο. Yes. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι το θέμα εδώ είναι η απαλλαγή της κοινοτικής υπηρεσίας ελέγχου της Ελίας. Προτού να, πω, να, προτού να περάσω στην ουσία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Διευθύντη της ε, Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της ελίας τον κύριο Μακέλ, που είναι και παρόν. Ε, ε επίσης ε, συνεργάστηκα ε, και με την ε, Επιτροπή ε, Ελέγχου του προπολογισμού και να ευχαριστήσω και, τη, και τον εκεί από την Γραμματεία. 11 εκατομμύρια ευρώ ήταν ο προϋπολογισμός Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλίας στις... και την προηγούμενη χρονιά σχεδόν το ίδιο 10 εκατομμύρια 600.000 ευρώ ε, διαπιστώσαμε ότι το εσωτερικό σύστημα ελέγχου των λογαριασμών, τον λογαριασμών λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να ε, τονίσουμε ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ε, το μοιράζεται με την ΕΜΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Αυτό είναι πολύ καλό, αποτελεί πολύ καλό παράδειγμα και για άλλους οργανισμούς. Κάποιες μικρές επικρίσεις βρήκαμε για Παράδειγμα, καθυστέρηση πληρωμών σε κάποιες μικρές περιπτώσεις, εξετάζονται οι λόγοι και μπορώ μόνο να επενέσω τον καλό και γρήγορο τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε μαζί μας ε, ε, ο οργανισμός αυτός. Ε, θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι έχει νέο όνομα. Δεν λέγεται πια CFCA, όχι κοινοτική υπηρεσία ελέγχου της Ελίας, αλλά ευρωπαϊκή EFCA ονομάζεται τώρα πια. Θα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό λοιπόν. Ο κύριος Ιαν Οσία ε, ε, από την Ιρλανδία ήταν ε, υπεύθυνο για το σύστημα ελέγχου. Ήταν πολύ καλές οι τεκμηριώσεις όλων των πληρωμών. Οι συναλλαγές ήταν νόμιμες και είχαν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον νόμο. Μια μικρή επίκριση. Δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη ο η αρχή ε, ε, του, του οικονομικού έτους, δηλαδή ε, χρήματα το 2010 χρησιμοποιήθηκαν το 2011, αυτό επιτρέπεται σε περιπτώσεις εξαιρετικές. Η, υπηρεσία έχει λάβει υπόψη σε αυτή τη, τη διόρθωση για το 2012. Έλειπαν κάποια στοιχεία και υπάρχει η σφραγίδα με ημερομηνία. Ε, ε, έτσι λοιπόν θα αποφευθούν ε, οι ελλείψεις ημερομηνιών στο παρελθόν. Επίσης όσον αφορά την επιλογή προσωπικού θα ήταν καλύτερο πριν την διαδικασία πρόσληψης να καθιερώνονται όλα τα κριτήρια. Αυτό θα γίνει και στο μέλλον. Το ελεκτικό συνέδριο είναι ικανοποιημένο με αυτές τις τροποποιήσεις. Παρόμοιε τροποποίησει θα γίνουν και σε άλλε υπηρεσίε. Αυτό λοιπόν δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Είναι σχετικά νέα αυτή η υπηρεσία. Από το 2005 και μετά υπάρχει και ε, διαπιστώνουμε ότι πολύ γρήγορα μαθαίνει από τα λάθη τη. Ε, Ω Επιτροπή έχουμε επισκεφθεί το Βίγκο που βρίσκεται η υπηρεσία αυτή και θα γίνει και περαιτέρω επίσκεψη ε, φέτος ε, τον Οκτώβριο. Ανοιχτή είναι η πόρτα της υπηρεσίας αυτής. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω στο Κοινοβούλιο την απαλλαγή της υπηρεσίας μας έπεισε η δουλειά τους και γνωρίζουμε ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ευχαριστώ πολύ. Μου έχεις δει το λόγο εκπρόσωπος του οργανισμού. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για ε, μια έκθεση που θεωρούμε πολύ θετική και ε, αντικατοπτρίζει την ε, εκτίμηση της δουλειάς μας ε, και αντικατοπτρίζει επίσης ε, τις πρόοδους που έχουμε σημειώσει όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο. Όσον αφορά την παραγραφό 4 θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όλες οι πολύ σημαντικές συστάσεις που, του, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου έχουν εξεταστεί και στον πιο πρόσφατο έλεγχο το, τα τέλη Οκτωβρίου. Όσον αφορά το σημείο 5 ε, τις παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι έχουμε υιοθετήσει αυτές τις παρατηρήσεις και τις έχουμε εφαρμόσει ε, Μικρές αλλαγές στην ε, διαδικασία μας ε, θα επιφέρουν αυτές τις παρατηρήσεις. Ε, τις έχουμε λάβει υπόψη μας. Μπορείτε να, ε, μπορώ να σας καθησυχάσω. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ. Muchas gracias. Ευχαριστώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι. Λοιπόν, η προθεσμία την κατάσταση τροπολογιών είναι για τις 27 Ιανουαρίου. Επίσης το μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι, 19, τροποποίηση του κανονισμού 1300-2008 για τη θέσπιση πολιτού σχεδίου του απόθυμα Ρέγκα που κατανάμε τα δυτικά τη Σκωτία για την ελεία του αυτού, κύριο Στίβενσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Συγγνώμη, ίσως να δώσουμε πρώτα το λόγο στην Κομισιόν. Μήπω θέλει να μας εξηγήσει κάτι ή να μας παρουσιάσει την πρόταση. Και κατόπιν ο εισηγητή. Παρακαλώ, από την Κομισιόν. Κύριε Φρίς. Thank you very um, Σας ευχαριστώ πολύ. Μπέρναρτ Φρύ, είμαι διευθυντής ε, υπεύθυνο στα πλαίσια της ε, DG Mare τα βασικά στοιχεία της πρότασης αυτής θέλω να σας παρουσιάσω αποτελεί μέρος με ενό γενικότερου εγχειρήματο να ευθυγραμμιστούν πολλές πράξεις συναπόφασης οι οποίες εγκρίθηκαν πριν την έγκριση συνθήκης της Λισαβόνας και που πρέπει ουσιαστικά να συμμορφωθούν περισσότερο με την ε, κατεξοδότηση πράξη που προβλέπονται στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις ε, πράξεις οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν, ένα κατάλογο συγκεκριμένο έχουμε και είδαμε ότι ο κανονισμός αυτός δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο, σε αυτή την επιστολή που έχουμε, αλλά εξετάζοντάς τον περαιτέρω είδαμε ότι και αυτός πρέπει με τη σειρά του να προσαρμοστεί. Είχε γίνει λοιπόν μια αρχική παράληψη την οποία τώρα διορθώνουμε. Η ε, πρόταση πολύ απλά περιλαμβάνει τρεις βασικές τροποποιήσεις ε, όσον αφορά τη διαχείριση του πολιτού σχεδίου διαχείρισης για το απόθεμα Ρέγκας. Έχει να κάνει με τροποποίηση του άρθρου 7, όπου στόχος εδώ πέρα είναι να καταφέρουμε να διαχειριστούμε τα αποθέματα Ρέγκας ε, παρέχοντας την μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ο στόχος ε, MSY φαίνεται στο άρθρο 3, όπου έχουμε συγκεκριμένε ε, αξίες όσον αφορά τη θνησιμότητα και την βιομάζα του αποθέματος. Οι αξίες αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, σε επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, η οποία θα πρέπει να προσαρμόζεται κάθε έτος. Το σχέδιο διαχείρισης βασιζόταν πλέον στο Συμβούλιο για να γίνει κάτι τέτοιο. Με τη συνθήκη τη Λισαβόνα δεν μπορεί να στοιχιστεί αυτό και γι' αυτό το λόγο προβλέπεται εξουσιοδότηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον για να γίνεται η προσαρμογή αυτή. Η δεύτερη τροποποίηση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να κάνει με το άρθρο 8, αναθεώρηση του σχεδίου μετά από την πάροδο κάποιων ετών. Στο παρελθόν εξοδότηση προς το Συμβούλιο δινόταν γι' αυτό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί η διάταξη αυτή με ό,τι προβλέπεται για τις νομοθετικές αυτές πράξεις, δηλαδή από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει την αξιολόγηση και συνέχεια μπορεί να κάνει μια πρόταση προς τους συνομοθέτες προκειμένου να τροποποιήσουν το σχέδιο αυτό, αν αυτό κρυθεί αναγκαίο. Η τρίτη τροποποίηση είναι καθαρά τεχνικής φύσης. Ουσιαστικά τροποποιεί τον τρόπο με τον οποίο ε, καλύπτεται μια περιοχή γεωγραφικά από αυτό το σχέδιο ε, διαχείρισης. Δεν θα περιλαμβάνεται πλέον στο βασικό άρθρο, το άρθρο 1, αλλά περιέρχεται στους κανονισμούς του κανονισμού, η οριοθέτηση της γεωγραφικής ζώνης. Αυτές είναι οι προτάσεις τροποποίησης, όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου, πρόκειται για μία απλώς πρόταση ανάμεσα σε πολλές άλλες, οι οποίες θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν στις ε, νέες διατάξεις, στις συνθήκη της Σαμπάνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε έχετε λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω βέβαια ένα-δύο προβληματάκια με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο στο οποίο αναφέρεστε βρίσκεται στα σπάργανα και από ό,τι φαίνεται έχει σταθεροποιήσει τα αποθέματα ρέγγας στα δυτικά της Σκοτίας. Το πρόβλημα είναι, εσείς είπατε ότι δεν θέλετε να έχετε πλέον γεωγραφικούς ορισμούς. Θέλετε πλέον το σχέδιο αυτό να καλύπτει το σύνολο της περιοχής 6α. Το συγκεκριμένο όμως σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε με την συνεργασία της ISIS και με το πελαγικό ΡΑΚ, αναφερόταν μόνο στο απόθεμα Ρέγκας στα δυτικά της Σκοτίας, 6α βόρειο τμήμα, ενώ προβλέπεται διαφορετικό σχέδιο για τη ζώνη 6α νότιο τμήμα. Να προσπαθήσετε τώρα να εφαρμόσετε εσείς τον κανονισμό αυτό σε δύο διαφορετικά αποθέματα, νομίζω θα προκαλέσει τεράστιο χάος και ουσιαστικά δεν θα είναι λειτουργικό στην πράξη το πρόγραμμα αυτό. Έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα εργασία, το οποίο έχει να κάνει μόνο με το 6α βόρειο τμήμα, απόθεμα Ρέγκα δυτικά τη Σκωτία. Αφήστε το έτσι. Μην αρχίζετε αυτή τη στιγμή να τον μπλέκετε, να τον μπλέχνετε με το νότιο τμήμα. Είπατε επίση ότι θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί το σχέδιο αυτό με τι συνθήκε τη Λισαβόνα. Και είπα ότι θα χρησιμοποιήσετε κατεξοδότηση αρμοδιότητε, ουσιαστικά αποκλείοντά μα εμά, του Ευρωβουλευτέ, από την όλη διαδικασία. Στο εφιστάμενο σχέδιο προβλέπεται απέτηση κάθε τέσσερα χρόνια να έρχεστε σε επαφή με το πελαγικό ρακ, να το συμβουλεύεστε, και εσείς από ό,τι φαίνεται το έχετε αποκλείσει αυτό, δεν το συμπεριλαμβάνετε πλέον στη νέα πρόταση. Επομένως δεν θα υπάρξει περαιτέρω τετραετής διαβούλευση, μετά την πάροδο τεσσάρων ετών μάλλον, χρησιμοποιείτε τις ε, κατεξοδότηση πράξεις και μόνο αν υπάρχει πρόβλημα μας δίνετε το δικαίωμα να επέμβουμε. Δεν το βρίσκω αυτό καθόλου ικανοποιητικό, λυπάμαι και θα υποβάλω μια τροποποίηση σχετική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκούν. Ως ε, σκιώδης εισηγητής ε, και μέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Στίβενσον, ε, μπορώ μόνο να συμφωνήσω μαζί του. Τα ε, πολιετή αυτά ε, προγράμματα διαχείρισης είναι πολύ σωστά ότι χρειάζονται επιστημονικά στοιχεία, ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τη θνησιμότητα, θα πρέπει να εξετάσουμε την βιομάζα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εμπειρίες των ΕΡΑΚ, των Περιφερειακών Συμβουλίων. Όπως όμως είπε ο κύριος Στίβενσον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τις διαφορετικές ε, συνθήκες ε, κάποιων περιοχών, όπως 6, 6α και 7. Γι' αυτό είναι σημαντικό εδώ στο Κοινοβούλιο να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και να μην τα αφήσουμε αποκλειστικά στο Συμβούλιο. Η πρόεδρος του Συμβουλίου από τη Δανία είπε ότι τα ΤΑΚ ε, χρειάζονται επιστημονικά ε, στοιχεία, ε, αλλά τα προγράμματα διαχείρισης συζητιώνται εδώ στο Κοινοβούλιο και αποτελούν σαν αντικείμενο στην απόφαση. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον κύριο Στίβενσον. Ευχαριστώ. Κομισιόν, παρακαλώ. Ναι. Μία διευκρίνηση να επιφέρω, αν το επιτρέπετε. Θα έπρεπε να το είχα πει αυτό στην αρχική μου ομιλία. Όσον αφορά την πρώτη παρατήρηση του εισηγητή, γεωγραφική κάλυψη. Κάνοντα την πρότασή μας, κάναμε ένα λάθο ουσιαστικά. Πρόθεσή μας δεν ήταν να διευρύνουμε τη γεωγραφική περιοχή. Πρόκειται για ένα τεχνικό σφάλμα που έχει γίνει στην πρόταση, θα το διορθώσουμε και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανταλλαγής επιστολών θα επέλθει η αλλαγή αυτή και ελπίζω ότι δεν θα γίνει αυτό πολύ αργά. Να διευκρινίσω λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε εμείς να διευρύνουμε το γεωγραφικό πεδίο. Μάλιστα, άλλο κανεί θέλει το λόγο. Όχι, ωραία, σα ευχαριστώ όλου. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε στι 3 ακριβώ το απόγευμα. Σα ευχαριστώ όλου.